Okay, welcome everybody. Καλώς ορίσατε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ορίζω τον Χωακίν Αλμούνια στην Επιτροπή μας. Δεν είναι ξένος, βέβαια. Θα συζητήσουμε τα περί ανταγωνισμού την τελευταία φορά. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψε με την Κομισιόν ε, και η ημερομηνία τότε έλεγε 27 Μαΐου. 8 Οκτωβρίου έπεται και η τρίτη σχετική συνεδρία, σας ε, το λέω από τώρα, αλλά στο μεταξύ μπορούμε να ακούσουμε τι θα μας πει ο Επίτροπος και ο συνήθως ε, να τεθούν και οι ερωτήσεις στη συνέχεια. Είναι εδώ οι περισσότεροι από την ομάδα εργασία για τον ανταγωνισμό από ό,τι βλέπω. Πρέπει να σας πω ποιοι είναι αυτοί βέβαια. Έχουμε να επανασυγκροτήσει αυτήν την ομάδα Αντολίνη Σάντσες Πρεσέδο είναι ο πρόεδρος. Uh, Αυτά είναι τα μέλη της ομάδας εργασίας που επεξεργάζονται την έκθεση ανταγωνισμού για φέτος. Μια ομάδα εργασία που επαναλαμβάνω επανασυγκροτήσαμε για το 2012. Ο Επίτροπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή Έκων και την Πρόεδρο, την κυρία Μπόουλς, που με προσκάλεσε να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση ανταγωνισμού για το 2011. Η σημερινή μας συνεδρίαση πράγματι λαμβάνει χώρα σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές, γενναίες αποφάσεις και πολιτική φιλοδοξία η έκβαση των ελληνικών κυριακάτικων εκλογών ήταν ένα θετικό βήμα και επιβεβαίωσε την θέση της χώρας στην Ευρωζώνη. Ένα άλλο σημαντικό βήμα όμως ε, το έχουμε μπροστά μας, σε δέκα ημέρες δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να λάβει αποφασιστικές αποστάσεις για να, αποφάσεις για να ε, επανεκκινήσει την χρηματοοικονομική οικονομική πολιτική ένωση το μέγεθος των προκλήσεων είναι η ηγεσία, πολιτική αποφασιστικότητα και ένα στρατηγικό όραμα. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού είναι ένα καθήκον πολύ σημαντικό που εδώ και ε, κάποια χρόνια και ιδίως από το 2008 και μετά με την κρίση έχει γίνει πολύ δύσκολο στόχος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αξιολογήσουμε επιτόπου ποιος είναι αντίκτυπος της κρίσης. Η έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα είναι ουσιαστικά η έκβαση αυτή τη εμπειρία. Και ο απότατο στόχο μα είναι να δημιουργήσουμε τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε για ανάπτυξη και απασχόληση στην εσωτερική αγορά. Πάνω από ποτέ είναι, περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό να βρούμε διέξοδο από την κρίση και να τονώσουμε την οικονομία και να απελευθερώσουμε βέβαια και το δυναμικό της ενέας αγοράς. είχε στήσει το Κοινοβούλιο να έχουμε μια νέα μορφή, δηλαδή ε, με βάση την πολιτική να ε, παρουσιάσουμε τα πράγματα στην έκθεση. Έχουμε λοιπόν τρεις τομείς, χρηματοοικονομικές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε, τρόφιμα και κρατικές ενισχύσεις. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας για εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύων είναι μια ανάπτυξη πολύ σημαντική στον τομέα της πολιτικής θέλω να την ε, συζητήσω σήμερα μαζί σας. Βέβαια δεν τη συμπεριλάβουμε στην έκθεση γιατί ξεκίνησε μόνο πριν από λίγες εβδομάδες. Αλλά καταρχάς θα σα πω κάποια πράγματα για τι χρηματοπιστωτικέ αγορές. Ο βασικός μας στόχο και το 2011 ήταν να διατηρήσουμε τη σταθερότητα παρά τις ε, αναταράξει και τι περιδινήσει συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε τις, ε, τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση διάσωση τραπεζών που χρειάζονταν δημόσια στήριξη για να έχουν την χρηματοπιστωτική του σταθερότητα. Θέλαμε να περιορίσουμε το κόστος για τις, δημόσιε για τις δημόσιες δαπάνες. Όταν όμως ε, δινώθηκε η κρίση του ε, δημόσιου χρέους, η μόνη επιλογή που είχαμε ήταν να επεκτείνουμε και να επιμηκύνουμε και το 2012 αυτό το καθεστώς για τις τράπεζες και θα έχουμε ένα νέο μόνιμο καθεστώς όταν σταθεροποιηθούν οι αγορές. Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να έχουμε νέε κατευθύνε γραμμέ ε, αναδιάρθρωσης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Υπό του ε, ειδικού κανόνες που εξακολουθούν να ισχύουν όπως είπα, αποφασίσαμε την βιωσιμότητα αναδιάρθρωση εκαθάριση 46 τραπεζών και εξεργαζόμαστε ακόμη το τι θα κάνουμε σε 25 περιπτώσει Για τέσσερα σχεδόν χρόνια Ήμασταν ε, και, αν θέλετε, μια αρχή διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας και τις ε, διαρθρωτικές κρίσεις, τα προβλήματα. Παρά όμως ε, του καλού μας ιστορικού, των καλού μας επιδόσεων, χρειαζόμαστε ένα πλήρες σύστημα διάσωσης και εποπτείας ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί λοιπόν με ένα ε, μηχανισμό εγγύηση των καταθέσεων έχουμε και κάποιες ιδέες σχετικά με την Τραπεζική Ένωση. Έτσι θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεσή τη και τα σωστά εργαλεία για την αποτελεσματική αναδιάρθρωση και διάσωση τραπεζών που θα έχει ω αποτέλεσμα να μην πληρώνει πλέον το λογαριασμό ο φορολογούμενο. Δεν περιοριζόμαστε όμω στη διαχείριση τη διάσωση των τραπεζών, τη δημόσια διάσωση των τραπεζών, αλλά έχουμε και κάποια θέματα αντιτράστ, αντιμονοπολιακά δηλαδή, που μα απασχολούν. Έχουμε δύο επιθέσει που αφορούν ε, υπερβολικέ τιμέ και περιορισμού ε, για ορισμένα δεδομένα ιδιοκτησιακά στι χρηματοπιστωτικέ οι αγορές. Η εταιρεία είναι η Standard Poor's, βρήκαμε κάποια λύση και έχουμε και ένα δεύτερο, μια δεύτερη υπόθεση, την Thomson Reuters. Τον Απρίλιο 2011 είχαμε δύο αντιμονοπολιακές υποθέσεις στην αγορά των CDS, των ασφαλιστρών κινδύνων, να δούμε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών τραπεζών που ίσως είχαν ε, υιοθετήσει στρατηγικές για να διατηρήσουν την ισχυρή τους θέση στην ε, αγορά, την επικερδή αγορά over the counter. Η υπόθεση τώρα CDS έχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που είναι η πρόσβαση στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Νομίζω ότι οι ανοιχτέ προσβάσιμε χρηματοπιστωτικέ υποδομέ είναι σημαντικέ για την παροχή αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε υπηρεσίε και επενδυτέ. Όπω γνωρίζετε από την πλευρά των συγχωνεύσεων, είμαστε υπέρ τη ανταγωνιστική ε, διάσταση, ε, συγκεκριμένα ε, στην απόφασή μα για την ε, για το γερμανικό χρηματιστήριο Euronext ε, Deutsche Börse Neise Euronext. Ένα άλλο τομέα στον οποίο είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι είναι οι αγορέ πληρωμών. Είχαμε την υπόθεση Mastercard πρόσφατα και η Δημιουργία των Ευρωπαϊκών Δικαστήριων επιβεβαίωσε τα πορίσματά μα ε, για τι πολυμερεί χρεώσει σε συνάλλαγμα. Και ε, για τη Visa θα, έχουμε, θα συνεχίσουμε τις έρευνες και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες ρυθμιστικές λύσεις για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου στον κλάδο αυτό. Νωρίτερα φέτος ξεκινήσαμε έρευνα ε, σε σχέση με τις πράξεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, διότι υπήρξαν κάποιοι ισχυρισμοί ότι τα πρότυπα διαλειτουργικότητας που ανέπτυσαν για τις γραμμικές πληρωμές θα δημιουργούσαν πολλά προβλήματα σε υπηρεσίες πληρωμών που προσφέρουν άλλοι ε, οργανισμοί και όχι τράπεζες. Επίσης υποστηρίζουμε την τυποποίηση για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ολοκλήρωση της αγοράς και βέβαια πρέπει να είναι δίκαιη και διαφανής η σχετική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να αποκλείσουμε καινοτόμου ε, outsiders. Έρχομαι στις αγορές τροφίμων. Από την πλευρά του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως αυτό που έκανε ήταν να αναθεωρεί ορισμένες διακρατικές συγχωνεύσεις ε, ευρωπαϊκής εμβέλειας. Για παράδειγμα, πρόσφατα ε, ολοκληρώσαμε την ε, απόκτηση με, ενός ε, μεγάλου εμπόρου ζάχαρης από την Σουντ Τσούκερ, το μεγαλύτερο παραγωγό ζάχαρη στην Ευρώπη με κάποια ένδικα μέσα που θα διατηρήσουν τον ανταγωνισμό στην Ιταλική αγορά. Επειδή όμω οι πολλέ αγορέ τροφίμων τείνουν να είναι είτε τοπικέ είτε εθνικέ, έχουμε συνεργασία με τι εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σε επίπεδο εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Βλέπουμε πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Ε, η ECN δημοσίευσε μία έκθεση τον προηγούμενο μήνα. Βλέπουμε ότι από το 2004 στο 2011 η Υπηρεσία της Ανταγωνισμού της Ευρώπης ε, διαχειρίστηκαν περίπου 1.300 υποθέσεις συγχώνευσης και 180 αντιμονοπολιακές υποθέσεις ε, με καρτέλ κατά το ίμιση που διασυλλογούν στον τομέα της επεξεργασίας μεταποίησης τροφίμων. Είδαμε διάφορα δομικά εμπόδια όπως ε, ρυθμιστικούς φραγμούς στις αγορές λιανικής πόλης σε κάποιες χώρες μέλη. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτά τα εμπόδια. Πέρυσι τον Δεκέμβριο εγκρίναμε επίσης ε, τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, γιατί περνάω τώρα στις πολιτικές εξελίξεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Το Μάρτιο αποφασίσαμε τα περί ε, των ταχυδρομείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν η πρώτη υπόθεση και πριν από ένα μήνα ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία εξυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων. Στόχο τη μεταρρύθμιση είναι να βοηθήσουμε τι κυβερνήσει, τι ευρωπαϊκέ, να προωθήσουν την ανάπτυξη όσο ταυτόχρονα βέβαια γίνονται και προσπάθειε δημοσιονομική εξυγίανση και προσαρμογή. Το καθεστώ που θα προκύψει από αυτή τη μεταρρύθμιση θα ενισχύσει ε, την ε, βοήθεια που θα στοχεύει κατά των αποτυχιών της αγοράς, θα προσφέρει πραγματικά κίνητρα, δεν θα δαπανά ούτε θα, θα διασπαθίζει τα χρήματα των φορολογουμένων. Καλή βοήθεια, δηλαδή που θα προσδοθεί και την περιβαλλοντική προστασία, θα στηρίζει την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία θα προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, αλλά μόνο όταν η στήριξη στηρίζεται, επαναλαμβάνω, σε γνήσιες αποτυχίες της αγοράς για να αλλάξει ουσιαστικά ε, τη συμπεριφορά των αποδεκτών. Αυτό που αντιθέτω θέλουμε να αποθαρρύνουμε τις κακές ενισχύσεις, κακή βοήθεια, δηλαδή διασπαθήσεις ε, που θα διατηρήσουν αναποτελεσματικέ αγορές στην αγορά. Και θα συγκεντρώσουν όλες ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Λαμβάνουμε υπόψη κατευθυντήριε γραμμέ για την περιφερειακή και εθνική βοήθεια, τι κατευθυντήριε γραμμέ για την ε, έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και τι περιβαλλοντικέ ενισχύσει. Τα δύο τρίτα περίπου των ποσών ε, αφορούν αυτά που σα προανέφερα. Τώρα η πρωτοβουλία επίσης ε, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ομαλό, ξεκάθαρο καθεστώ με αλλαγέ που θα περιλαμβάνουν επικαιροποίηση του κανονισμού, αναθεώρηση των κανονισμών General Block Exemption και Enabling Regulation ή και του κανονισμού περί ελαχίστων, de minimis regulation. Θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις που έχουμε, τις αποφάσεις που θα εγκρίνουμε και για τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες. Φέτος, νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να στείλουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις αλλαγές στους διαδικαστικούς κανονισμούς των Procedure και Enabling Regulation. Θέλω να σας ενημερώσω και θα σας ενημερώνω σε τακτά διαστήματα για τις προτάσεις που θα διατυπώσουμε για τροποποίηση σε οποιοδήποτε άλλο κανονισμό, τομεκέ, περιφερειακέ κατευθυντήριες, γραμμές, έρευνα, ε, επιχειρηματικό κίνδυνο, κεφάλαια, περιβαλλοντική βοήθεια κτλ. Όλα αυτά, ό,τι σας ενδιαφέρει, θα μπορούμε να το συζητούμε είτε ε, ε, με τη δική μου παρουσία είτε με μέλη τη δική μου ομάδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό που θα σας έλεγα να κάνουμε τώρα, να περάσουμε στις ομάδες εργασίας, αυτές που ετοίμασαν τις εκθέσεις πρωτοβουλίας, θα περάσουμε σε αυτούς λοιπόν. Άντολη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ως εισηγητής για την επόμενη έκθεση ανταγωνισμού, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί διατηρεί διάλογο με την ομάδα εργασία ε, τη Επιτροπή μα ε, στο θέμα πάντα του ανταγωνισμού και γιατί είναι πολύ συνεργάτησιμο μαζί μα. Η έκθεση, είπατε ότι είναι μια νέα μορφή ε, που υιοθετείται σε αυτή την έκθεση και πράγματι η έκθεση περιλαμβάνει τα θέματα που μα έχουν απασχολήσει στην ομάδα εργασία. Τρει βασικοί άξονε, σημαντικοί για μα. Πρώτο, η συμβολή τη πολιτική ανταγωνισμού στην αντιμετώπιση τη κρίση που βιώνουμε. Δεύτερο άξονα. Πώ μπορεί η πολιτική ανταγωνισμού να συμβάλλει και αυτή ε, στη διέξοδο από την κρίση και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, ανάπτυξη και απασχόληση δηλαδή. Τρίτος άξονας, διάλογος με άλλα θεσμικά όργανα, διάλογος και συνεργασία μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Αυτές λοιπόν οι τρεις γραμμές ε, που μας απασχολούν, οι τρεις άξονες ε, εργασίας. και εκεί επικεντρώνεται και συστάση που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να εστιάσω εγώ στην κρίση, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο επίκαιρο και επίγον ζήτημα. Έχει αποδειχθεί ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, διατήρηση της διαφάνειας των αγορών και του θεμητού, του δίκαιου ανταγωνισμού. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν την ενεργοποίηση προγραμμάτων επανακεφαλαιοποίησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανακεφαλαιοποίησης ε, ευρωπαϊκών ε, ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Θέλω να σας θέσω σχετικά λοιπόν τρία ερωτήματα κύριε Επιτροπέ. Πρώτον, οι κανόνες που εφαρμόζονται μέχρι τώρα μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ή απαιτούνται νέοι κανόνες. Δεύτερο ερώτημα. Από πλευρά ανταγωνισμού υπάρχει κάποια διαφορά αν γίνει άμεσα ε, η επανακεφαλαιοποίηση ή μέσω των κρατών μελών. Υπάρχει διαφορά ε, από το ένα στο άλλο. Και τρίτο ερώτημα. Αυτή η επανακεφαλαιοποίηση εξυγένωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα λάβει υπόψη τον ηθικό κίνδυνο, θα προστατεύσει τους ε, φορολογουμένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντσεθ Πρεσέδο και για το έργο το οποίο επιτελείται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τον ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ για τις εργασίες και τη δική σας εργασία ως εισηγητού για την εκπόνηση επόμενης έκθεσης της ετήσιας έκθεσης, πάνω στην ετήσια μάλλον έκθεση, της ε, γενικής δομές σας παρουσίασα. Θα απαντήσω όμως απευθείας στα συγκεκριμένα σας ερωτήματα. Οι κανόνες που θα ισχύσουν στο μέλλον, δεν μπορώ να σας δώσω μια ε, οριστική όμως αυτή τη στιγμή ημερομηνία, είναι αυτοί οι οποίοι τώρα ισχύουν. Δεν ξέρω αν όπως είχαμε κάνει στα τέλη του 2010 ή 2011, ε, δεν ξέρω μήπως χρειαστεί κάποια μικρή ε, προσαρμογή. Αλλά οι κανόνες κατά βάση θα είναι το ίδιο. Έλεγχο κρατικών ενισχύσεων με το πιστοτικό σύστημα. Οι κανόνε ίσχυσαν τέλη 8, αρχέ 9. Τέσσερα είναι τα βασικά κείμενα για την επανακεφαλαιοποίηση, για την αντιμετώπιση κάποιων τοξικών προϊόντων, για τις εγγύσεις, ε, δημόσιες εγγύσεις και για την αναδιάρθρωση των κρατικών ιδρυμάτων. Αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι ότου ομαλοποιηθεί κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι για να σας παρουσιάσουμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, τους νέους δοσανατολισμούς για τη διάσωση και αναδιάρθρωση χρηματοπιστωτικών ε, οντοτήτων, αλλά σε κανονικές ε, συνθήκες, σε ομαλές συνθήκες, αν μου επιτρέπετε. Όμως βλέπουμε ότι η κρίση, επειδή θα διαρκέσει δυστυχώς ακόμα μήνες, ίσως και χρόνια, δεν ξέρω, δεν νομίζω δυστυχώς ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα ομαλό καθεστώς. Είμαστε ακόμα σε ένα καθεστώς αντιμετώπισης ε, έκτακτης ανάγκης, ένα ε, καθεστώς για αντιμετώπιση της κρίσης είναι διαφορετικό ε, το αν θα γίνει επανακεφαλοποίηση με εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια από τα κονδύλια της Ευρωζώνης. Αν θα γίνει με τα κράτη-μέλη διαφορετικό, αν χρησιμοποιηθεί δηλαδή ο νέος μηχανισμός και διαφορετικά θα είναι αν χρησιμοποιηθεί άμεσα με τα bank stops, τις τράπεζες. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι οι οριζόντιες συνθήκες ουσιαστικά, όχι ο έλεγχος. Ο έλεγχο είναι ο ίδιο. Σε ό,τι αφορά τον ηθικό κίνδυνο, είναι προφανές ότι υπάρχει. Όποτε χρησιμοποιούμε δημόσια ε, χρήματα, δημόσιους πόρου για να στηρίξουμε κάποιες επιχειρήσεις, κάποιους φορείς και όχι κάποιες άλλες ε, εταιρείε υπάρχει ηθικός κίνδυνο τον οποίο προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε στο βαθμό και στο μέτρο του δυνατού. Ο ηθικός κίνδυνος υπολοιματικό, αν θέλετε, που δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε εντελώ, θα αντισταθμιστεί από τα ωφέλη που θα προκύψουν λόγω τη χρηματοπιστωτική και χρηματοοικονομικής σταθερότητα και την αποφυγή των συστημικών κινδύνων. Πώ μπορούμε να αποφύγουμε τον ηθικό κίνδυνο με τη συζήτηση, με το διάλογο που πολλέ φορέ είναι δύσκολη συζήτηση για τα σχέδια αναδιάρθρωση και τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα πρέπει να προκύψουν. Δεύτερο, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον ηθικό κίνδυνο πάλι με τη συζήτηση, πάλι δύσκολη ενίοτε, της κατανομής προσπαθειών και ε, μεταξύ των ομολόγων, ε, των μετόχων, δημοσίων αρχών κτλ. Και τρίτον, προσπαθούμε να εξαλείψουμε αν μπορούμε τη, δια, ε, τη στρέβλωση ανταγωνισμού. Δηλαδή κάποιες που έχουν ε, πάρει βοήθεια ε, να υποστηριχθούν τελικά αθέμητα, ενώ άλλες οι οποίες δεν έχουν λάβει βοήθεια αντιμετωπίζουν τελικά προβλήματα στις αγορές. Ε, ευχαριστώ. Ο περσινός πρόεδρος, κύριος Σφαμπ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο. Ε, είχετε αναφέρει ότι ε, αυτό είναι ένα θέμα που είναι δύσκολο και έχει και πολιτικό προσανατολισμό. Είπε ο συγγετής ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την άλλη. Νομίζω το κοινοβούλιο θα πρέπει λίγο να μην είναι ικανοποιημένο γιατί όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε και τα οποία έχουν υιοθετηθεί δεν βρίσκονται στη νέα έκθεση. Αλλά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και γι' αυτό χαίρομαι που είμαστε εδώ. Το πρώτο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι όπως και πάντα ε, σκέφτομαι ε, εάν ε, υπάρχει δυνατότητα η Κομισιόν στον κανονισμό 1 του 2003 σχετικά με τα πρόστιμα ε, να ε, ενσωματώσει αυτά τα νομικά εργαλεία. Υπάρχει ένας, ένα πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτό. Απ' την άλλη θα ήθελα να συγχαρώ γιατί κάνατε αυτό που είχατε πει το 2009. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, non-product businesses, ε, προωθούνται και ειδικότερα αυτές που έχουν συγκεκριμένα ε, προϊόντα ε, ενώ τα καρτέλ τιμωρούνται. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό που έχουν μειωθεί και τα παράθυρα και χαίρομαι ε, για το γεγονός ε, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα συμμορφώνονται και αυτές στο μέλλον με τις γραμμές της Κομισιόν Τρίτων. Ήθελα να ρωτήσω σε τι βαθμό συζητά η Κομισιόν για την μέτρηση του ύψους ενός προστίμου, δηλαδή ε, θα μπορούσε να γίνει μια διαιτησία μεταξύ αυτών που παραβαίνουν τον ανταγωνισμό και αυτών που πλήττονται από τα καρτέλ. Ίσως ε, αυτοί που θα πάρουν ε, τα χρήματα θα πρέπει να έχουν κάποια να, να τηρούν κάποιους κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σφάμπ. Να σας απαντήσω στα δύο ερωτήματα που θέσατε. Πρώτον, τα πρόστιμα. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή σα, αλλά με τον κύριο Σφάμπ επίση το έχουμε συζητήσει επαλημένω και διμερός. Η συγκεκριμένη ε, περίπτωση, τα mounting windows που αναφέρατε, δείχνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε ό,τι θέλουμε ουσιαστικά με τα πρόστιμα είστε νομοθετικό σώμα, σας αρέσει να νομοθετείτε και εμένα, ε, όταν είμαι βουλευτή. Αλλά πρέπει να ορίζουμε τις προτεραιότητες και αυτό σε συνάρτηση με τους στόχους και τις ανάγκες. Οι στόχοι που επιδιώκουμε με την πολιτική μας για τα πρόστιμα που επιβάλλουμε ε, σε διάφορα καρτέλ, ε, σε περιπτώσεις που έχουμε μονοπωλιακές καταστάσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 6 μήνες βέβαια, αλλά ε, ίσως μου πει ε, κάτι ότι χρειάζεται να αναθεωρηθεί αυτός ο κανονισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια άποψη. Νομίζω ότι με βάση τους κανόνες που έχουμε, το νομικό πλαίσιο που ισχύει, τα πρόστιμα αποδίδουν τα αναμενόμενα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συμφωνίες. Από το 2010 έως ε, τούδε έχουμε υιοθετήσει διάφορες συμφωνίες διακανονισμού, settlement και σε καρτέλ και ε, σε αντιμονοπολιακά ε, ζητήματα. Σε περίπτωση καρτέλ διάφορες ε, υποθέσεις. Ε, το 11 νομίζω τέσσερις υποθέσεις είχαμε με διακανονισμό. Και όσες επιχειρήσεις ε, λαμβάνουν μέρος στους διακανονισμούς, εκεί μειώνεται το πρόστιμο κατά 10%. Τώρα, στην περίπτωση ε, έχουμε το άρθρο 9 του κανονισμού. Έχει γίνει με την IBM, με άλλες υποθέσεις και με την Google που το πρότεινα και περίμενα την απάντησή τους ή Standard Poor's που σας προανέφερα. Αν η εκάστοτε εταιρεία θέλει να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο, τη διαδικασία των commitments με βάση ε, το άρθρο 90 μπορούμε να έχουμε αυτή τη διαδικασία για τις διάφορες δεσμεύσεις. Μπορούν λοιπόν τα καρτέλ και τα τραστ να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να διερευνούμε την υπόθεση ε, για να δούμε αν υπήρξε παραβίαση ή όχι. Απλά δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε εταιρείε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό που κάνω είναι να ε, καλώ τα μέλη από την ομάδα εργασίας πρώτα και μετά όσοι άλλοι μου, ναι, μου γνέψουν. Ε, φαντάζομαι ότι όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας θέλουν να μιλήσουν. Ε, Γκούνα, Σόφι, Φίλιπ, μετά, Ντέρκεν και Γιώργεν. Και μετά ήδη στη λίστα μου έχουν το τα τα Edward Cicluna, Roddy Kretzer and myself. And Diogo Feo. Anybody else going to wave? Well, we'll take... Είναι κανένας άλλος που θέλει, θα το πείτε στη... όσο προχωράμε. Γκούνα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την έκθεση ανταγωνισμού, κύριε Επίτροπε. Σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπάρχει ανάγκη να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι αποτελούν τεράστιο κόστος για τα κράτη-μέλη. Και σε χρο... καιρούς που χρειαζόμαστε να προσέχουμε, είναι σημαντικό να προσέχουμε και ε, αυτή την ε, οπτική γωνία των κρατικών ενισχύσεων. Νομίζω επίσης ότι θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει μια παρακολούθηση, ένα follow-up ε, το, του πώς οι κρατικές ενισχύσεις σε διάφορους τομείς, τον τραπεζικό τομέα κτλ. Ε, βοήθησαν στην επίτευξη στόχων. Μπορεί να υπάρχει εξ αρχή μια αξιολόγηση επιπτώσεων, αλλά πρέπει να υπάρχει και εκ των υστέρων μια παρακολούθηση για να δούμε εάν τα πράγματα πήγαν όπως είχαμε ε, υπολογίσει. Σχετικά με τις υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε από την Κομισιόν τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε δημόσιες επιχορηγήσεις σε διάφορες υπηρεσίες οικονομικού ε, ενδιαφέροντος, ε, αυτές ε, υποστηρίζουν τον τελικό χρήστη, τους καταναλωτές και όχι τις εταιρείε. Γιατί σε αυτούς τους τομείς είναι σημαντικό να υπάρχει πλουραλισμός και ανταγωνισμός και ανάπτυξη. Ο στόχος δεν είναι να υποστηρίξουμε τις εταιρείε αλλά τους πολίτες και θα ήθελα να ακούσω από εσά αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι να το αναπτύξουμε αυτό περαιτέρω. Διότι οι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο αποτελούν ένα τεράστιο κομμάτι του τομέα των υπηρεσιών που χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό. Σχετικά με κάποια άλλα θέματα που θέλω να θίξω. Ένα από τα πιο σημαντικά ίσως είναι το γεγονός ότι κάποιες φορές σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο εταιριών υπάρχουν διάφοροι φραγμοί εισόδου ε, που γύρονται για τις νέες εταιρείε. Βλέπουμε κάποιες κατατάξεις. Ας πούμε, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει τη δική της κατάταξη σχετικά με το που μπορεί κανείς να επιχειρήσει. Και είναι σημαντικό ε, ε, γιατί εξηγεί ε, γιατί έχουμε λήψη ανάπτυξη, ε, λίγη καινοτομία, λίγε επενδύσει και νέε θέσει εργασία. Θα ήθελα να ακούσω από εσά ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε και αυτή την πτυχή της πολιτικής ανταγωνισμού επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόμουερ. Σχετικά με την παρακολούθηση, το follow-up των κρατικών επιχορηγήσεων ποιες είναι οι επιπτώσεις και τα ωφέλη αυτών. Έχουμε περιορισμένους πόρους φυσικά, αλλά ένα από τα στοιχεία αυτού του πακέτου συγχρονισμού που ανέφερα στην αρχική μου παρουσίαση είναι να επιτρέψει μια καλύτερη ανακατανομή των πόρων μας με έμφαση στις ε, περιπτώσεις ε, που ε, εξάντεκ των ξέρουμε ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και επίσης ε, και ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον έλεγχο των εξαγωγών. Έχει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τέτοια ε, παρακολούθηση σχετικά με αξιολόγηση εκ των υστέρων των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν στο παρελθόν. Όσα συμπεράσματα έχουν βγει ως τώρα δείχνουν ότι το ποσοστό προβληματικών περιπτώσεων, όπου δόθηκαν δηλαδή κρατικές ενισχύσεις με βάση εθνικά σχέδια, τώρα εκ των υστέρων ε, αποδεικνύονται ε, και τώρα το, εκ των υστέρων αποδεικνύονται προβληματικά είναι γύρω στο 40%. Άρα υπάρχει συνυπευθυνότητα των κρατών μελών όταν συντάσσουν αυτά τα σχέδια που επιτρέπουν στις εταιρείε να επιχορηγούνται και όταν παρακολουθούν, εφόσον έχει ληφθεί ε, ε, θετική απόφαση, ε, όταν παρακολουθούν πώς λειτουργούν αυτές οι επιχορηγήσεις. Νομίζω ότι είναι μια κοινή ευθύνη. Η άδεια για την παροχή κρατικής ενίσχυσης είναι αποκλειστική ευθύνη της Κομισιόν. Το να προσέχει κανείς τι συμβαίνει μετά την θετική αυτή απάντηση είναι ε, θέμα συνυπευθυνότητας. Δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε όλα, όλες τις προϋποθέσεις ε, ε, για να έχουμε μια επιτυχημένη παρακολούθηση εκ των υστέρων χωρίς όλα αυτά. Για τις υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος, πέρυσι υιοθετήσαμε κανόνες, ένα πλαίσιο που είναι πολύ καλό όχι γιατί το έκαναν οι φίλοι μου από την Κομισιόν, αλλά γιατί πραγματικά έχει βελτιώσει ε, την εμπειρία μας ε, μετά από το πακέτο του 2005. Και ένα από τα στοιχεία αυτού του νέου πλαισίου είναι ότι δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι στο παρελθόν στο τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο αποτελεσματικότητας ε, όταν η εταιρεία που έχει λάβει τις επιχορηγήσεις χρησιμοποιεί τα χρήματα που έλαβε για να, παράσχει, να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος ε, των δημόσιων υπηρεσιών. Ε, ε, δεν είναι να πληρώσουμε μόνο τις εταιρείε για να ξεστα... αντισταθμίσουμε την προσπάθεια που κάνουν για να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, αλλά να... είναι για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Θεωρώ ότι θα πρέπει, ε, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη στόχο της, της πολιτικής ανταγωνισμού που είναι κατά των φραγμών στην είσοδο ε, και τη δημιουργία ε, ίσων ευκαιριών με έλεγχο των καρτέλ, έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και των αποφάσεων συγχωνεύσεων ε, και αντιτράστα αποφάσεις. Όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι φραγμοί μπορεί να υπάρχουν παντού, αλλά ειδικότερα πρέπει να προσέχουμε και προσέχουμε τις ε, βιομηχανίες δικτύου, όπου υπήρχαν κρατικά μονοπόλια και συνεχίζουν να υπάρχουν και πολλές φορές προσέχουμε ε, και τις νέες ε, δραστηριότητες, ε, νέες πατέντες, νέες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί χάρη στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Όλα αυτά δημιουργούν ευκαιρίες κατάχρησης εξουσίας και γι' αυτό πρέπει να εξισορροπήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Να είναι μια προσέγγιση η οποία θα ελέγχει αλλά δεν θα παραλύει και την καινοτομία. Γι' αυτό ήθελα ε, ένα κομμάτι της ε, παρουσίας μου εδώ ε, να το αφιερώναμε σε αυτό το θέμα. Θα το ήθελα πολύ γιατί είναι σημαντικό, γιατί δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες που υπάρχουν με την έναρξη που υπήρχαν με την έναρξη αυτού του τεράστιου ευρωπαϊκού ε, έργου πριν από 20 χρόνια. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Σόφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για τις ε, κρατικές ενισχύσεις, αλλά μετά άκουσα τα όσα είχατε να πείτε. Ελπίζω να μην κατάλαβα καλά ε, ότι αποδεικνύεται ότι το 40% των κρατικών ενισχύσεων είναι προβληματικό. πέστε μου ότι κατάλαβα λάθος. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τους ε, Διάφορου διάφορους, μύθους που κυκλοφορούν ε, δεν ξέρω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει η Επιτροπή τώρα, αργότερα. Το τρίτο ερώτημα. Το Κοινοβούλιο στις αιτήσεις εκθέσεις για τις Επιτροπές Ανταγωνισμού ζήτησε να γίνουν έρευνες στις μηχανές αναζήτησης και στις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Έγινε η έρευνα για το Google και είπατε ότι αυτό καλύπτει τις, αυτό που ζητήσαμε. Τώρα γνωρίζουμε ποια είναι τα προτινόμενα αντίδοτα από την Επιτροπή δεν ε, είναι ικανοποιητικά κατά τη γνώμη μου και δίνουν την εντύπωση ότι μάλλον μπορούμε να φανταστούμε το αποτέλεσμα. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εδώ. Οι διάφοροι τομείς αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς. Σιγά σιγά αρχίζουμε, <clears throat> αρχίζουμε να διαμορφώνουμε μια καλύτερη ιδέα των ποσών που παίζονται και του ανταγωνισμού Μήπως θα πρέπει να αντιδράσουμε εκ των προτέρων, να παρέμβουμε περισσότερο. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για μια αγορά θύλακα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με κυρίαρχους παίκτες. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να δράσουμε εκ των προτέρων και να κάνουμε κάτι αντί να περιμένουμε μέχρι που οι μεμονωμένες περιπτώσεις ή διάφορες διαμαρτυρίες φτάσουν μέχρι την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη απάντηση καταλάβατε πολύ καλά. 40% των περιπτώσεων, όχι του ποσού των κρατικών ενισχύσεων, των περιπτώσεων που αναλύσαμε σαν αποτέλεσμα μιας διαρκούς άσκησης ελέγχου ως προς το πόσοι χώρες, χώρες μέλη χρησιμοποιούν τον κανονισμό των εξαιρέσεων φαίνεται ότι το 40% των περιπτώσεων είναι προβληματικές. Μιλάμε για θέματα καθάρισης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Δεύτερον, ΚΑΤ. Δεν ξέρω αν το διάβασα αυτό το κομμάτι και σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη φορά που το πω δημοσίω. Νομίζω ότι αξίζει το λόγο, τον ε, κόπο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ρύθμιση στον τομέα το ΚΑΤ. Στο Ηνωμένο, στις Ηνωμένε Πολιτείε το έκαναν όταν ε, υιοθέτησαν την νομοθεσία Dotrang. Εμείς έχουμε να κάνουμε με αυτά τα ποσά από την άποψη ε, τη, του αντιτράστα, μιλάμε για τη Mastercard, μιλάμε για την ε, Visa. Δεν είναι άμεση η ευθύνη μου. Καταλαβαίνω τα όσα λέει ο κύριος Μπαρνιέ για τις κάρτες, για τις πιστοτικές κάρτες. Θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας ε, με τον κύριο Μπαρνιέ, με όλη την Επιτροπή, αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να προωθήσουμε κάποια νομοθεσία. Γιατί έχουμε να κάνουμε διαρκώς με περιπτώσεις που εφεσιβάλλουν στο δικαστήριο, που παίρνει αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Mastercard, για τη Visa. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει η ιστορία με τη Visa. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα συζητάμε ε, πέρα από τα πλαίσια του τομέα των πισωτικών καρτών. Μιλάμε για το ε, ε, σύστημα online πληρωμών. Έχουμε δημοσιεύσει μια πράσινη βίβλο, ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις, συζητάμε τώρα για να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με όλες αυτές τις ιδέες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν αποκλείω επουδενή το να υπάρξει κανονισμός. Αλλά βεβαίως δεν είμαι μόνος μου που θα μπορούσα να υιοθετήσω αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μηχανές αναζήτησης, τους τομείς αναζήτησης, το Google έχει το 90% των μηχανών αναζήτηση εδώ στην Ευρώπη και έχουμε να κάνουμε με το Google. Έχουμε, έχουμε επιληφθεί με την ε, περίπτωση που ε, πυροδότησε την ε, συγγραφή αυτής της επιστολής της κυρίας Σμιθ και περιμένω την απάντηση. Δεν, ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αν θα ακολουθηθεί η συνήθιση διαδικασία αντιτράστα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, την περίπτωση Google, η αντίρρηση υπαριθμών 1 που στείλαμε στην Google αναφέρεται στην κάθετη έρευνα, ε, στην κάθετη αναζήτηση. Οι περισσότεροι παίκτε στον τομέα της αναζήτησης αποτελούν μέρος αυτής της συζήτησης. Όχι ω δυνητικοί παραβάτες, αλλά ως δυνητικά θύματα της παραβίασης αυτή. Έχουμε, να, ε, ε, ε, έχουμε επιληθεί αυτού του τομέα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε να κάνουμε με την Google. Είναι η πρώτη φορά που έχει ξεκινήσει μια επίσημη ε, ανάκριση, μια επίσημη έρευνα. Για παράδειγμα όμως, μερικά θέματα που βασίζονται σε μερικές διαπαρτηρίες που αφορούν το Android, το λειτουργικό σύστημα δηλαδή της Google, ε, βρίσκονται σε φάση ανάλυσης από τις υπηρεσίες μου. Πιστεύω ότι δεν μιλάμε μόνο για την έρευνα που γίνεται σε ένα τομέα, μιλάμε για κάτι ευρύτερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Γαλλικά ή αγγλικά, τι προτιμάτε. Όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, τρία ε, σημεία. Θα ήθελα να αναφερθώ στις κρατικές ενισχύσει στο τραπεζικό τομέα. Για μένα, δεν ξέρω αν θα το γνωρίσετε δημοσίως, αλλά ε, έχουμε απασχολήσει πολύ το δικό σας τομέα σε ό,τι αφορά ε, τις ε, τράπεζες. Ποια είναι τα μαθήματα, που, ποια είναι τα διδάγματα που έχουμε μάθει από τις περιπτώσεις ε, που έχετε αναλάβει μέχρι τώρα και κυρίως ε, ποια είναι... Ποια είναι τα διδάγματα από το παρελθόν και πέστε μου αυτά τα παθήματα, μαθήματα σας ε, οδηγούν στο να υιοθετήσετε μια πιο αυστηρή στάση. Αυτό που θέλω να πω ότι μέχρι τώρα αφήσαμε ε, να ε, βιώνουν ε, οργανώσεις πραγματικά που ήταν τιμοθάνατες ε, με τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι στο χρηματοπιστωτικό ορίζοντα υπάρχουν ε, πολλοί φορεί που δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι κρατικές ενισχύσει. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι για μας ε, ορισμένα θέματα φορολογικού ανταγωνισμού ε, συνδέονται άμεσα με εκτροπές στην αγορά. Σας ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα αυτό, σας ενδιαφέρουν οι φορολογικές πρακτικές που θα μπορούσατε να θεωρήσετε και ως κρατική ενίσχυση σε ορισμένες επιχειρήσεις. Και τελευταίο σημείο, εδώ αναφερθήκατε, αναφερθήκαμε σε μία περίπτωση χειραγώγησης του Λιμπούρ. Θα ήθελα να γνωρίσω από αυτή την άποψη αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ευχαριστώ. Merci, merci, Ευχαριστώ. Καταρχά οι τράπεζες το σύστημα ελέγχου των τραπεζών, του, με των κρατικών ισχύσεων στις τράπεζες. Δεν ξέρω αν είχατε έρθει στην αρχή της παρουσίασής μου, εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Χρησιμοποιούμε τον έλεγχο, τα εργαλεία που έχουμε εμείς ως Επιτροπή για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων ως ένα σύστημα ε, εξυγίανσης de facto των τραπεζών. Έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα ε, γιούρ, ένα σύστημα ε, αντιμετώπισης της κρίσης. Δεν είναι ένα από τα στοιχεία που αφορούν την Ένωση Τραπεζών. Θυμάμαι τα επιχειρήματα που άκουσα όταν είχα ένα άλλο χαρτοφυλάχιο και αυτά ήταν θέματα που άκουγα κάθε ε, μήνα. Από ό,τι φαίνεται προχωράμε μέσα αυτό το τομέα, επιτέλους. Όσο δεν έχουμε μία αρχή εξυγίασης, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα, τα οποία έχουν τα ωριά τους. Αναφέρεται την τέξια. Βρισκόμαστε στη δεύτερη συζήτηση την τέξια. Η πρώτη, πρώτη απόφαση υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2010 Μόλις δηλαδή είχα αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, υπήρξαν δυσκολίες για την εφαρμογή του προγράμματος. Όλα αυτά αναφέρθηκαν από την Επιτροπή στην απόφαση του Φεβρουαρίου. Μετά το κρατικό χρέος δημιούργησε επιπρόθεστα ε, προβλήματα και τώρα όπως το γνωρίζετε είμαστε σε φάση ανάλυσης μιας απόλυσης ενός μέλους της Δέξια στην τράπεζα του Λουξεμβούργου σε μια τρίτη χώρα, σε ένα χρησιμοποιητικό ή ε, μια τρίτη χώρα. Εξετάζουμε το ε, θέμα της αναδιάρθρωσης της ΔΕΞΗ, η οποία έχει ε, κρατικοποιηθεί από το βελικό κράτος και είμαστε σε φάση αναδιάρθρωσης ε, για το σύνολο του ομίλου και για την ΔΕΞΗ ακριτή λοκάλα χρειάστηκε να περιμένουμε λίγο γιατί λόγω της διεξαγωγής των εκλογών στη Γαλλία τώρα με τη νέα κυβέρνηση στη Γαλλία, με την βελγική κυβέρνηση αυτή είναι η βασική ε, μέτοχη παράλληλα με τις αρχές του Λουξεμβούργου θα ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση πάνω σε μια επικοδομητική, περισσότερο θετική βάση. Βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα. Ε, προσωρινά χρειάστηκε να ε, χρησιμοποιήσουμε κρατικές εγγύησεις που είναι απαραίτητες. Όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και αλλού, ιδιαίτερα όμως στη Γαλλία επιμένω. Μόλις εσείς ως Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθετήσετε επιτέλους την ε, ε, οδηγία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εξυγίασης, εγώ θα είμαι περισσότερο ε, Ήσυχο, περισσότερο ήρεμο, όχι μόνο ως επίτροπος αλλά και ω ευρωπαίο πολίτη. Γιατί χρειάζεται μια τέτοια, χρειάζεται ένα τέτοιο φορέα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα συστήματα, θα πρέπει να σα πω στην εφαρμογή των προγραμμάτων που υιοθετήθηκαν από την εφαρμογή, Επιτροπή, η περίπτωση της Δέξια ήταν η πιο δύσκολη και συνεχίζει να είναι η πιο δύσκολη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ενός προγράμματος, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, πήραμε πολλές αποφάσει. Ε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι αποφάσεις εφαρμόζονται καλά με, με διαφορά χιλιοστών από την αρχική απόφαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα εδώ στο Βέλγιο διαπραγματευτήκαμε την ε, αλλαγή ενός αντίδοτου ε, ε μίας λύσης ε, για μια άλλη λύση ισοδύναμη. Εργαζόμαστε και στις τρεις χώρες της ζώνης του ευρώ με ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, Ευρωπαϊκή Ένωση Νομισματικό Ταμείο, επί του συνόλου του ε, τραπεζικού συστήματος και αυτό στην ε, Ελλάδα, την ε, Πορτογαλία και στην Ιρλανδία και στην Ισπανία θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Υιοθετήθηκε την περσμένη εβδομάδα ένα πρόγραμμα από το Eurogroup κατόπιν αιτήματο τη Ισπανία και ελπίζω ότι θα είναι έτοιμο τι επόμενε μέρε. Και σε γενικέ γραμμέ. Θα έλεγα ότι οι άλλε περιπτώσει δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα από την άποψη των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν ορισμένε περιπτώσει πιο δύσκολε. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στο Landesbank της Βαβαρίας, όπου δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και σε γενικές γραμμές. Τα πάμε αρκετά καλά με τις αρχές των χωρών που έχουν ακόμα προβλήματα προς επίλυση σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των φόρων και των κρατικών ισχύσεων υπάρχουν ορισμένα όρια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ω εκτροπή του ανταγωνισμού το γεγονό ότι μια χώρα μέλο καθορίζει ένα ποσοστό ε, φορολόγηση των εταιριών πιο χαμηλό από την γειτονική χώρα. Η συνθήκη δεν μα επιτρέπει να το θεωρήσουμε εκτροπή του ανταγωνισμού. Αλλά Μα απασχολούν όλες αυτές οι φορολογικέ ε, περιπτώσεις. Μόλι ε, του τους μήνε, μήνες ε, συζήτησα με την Ιταλική κυβέρνηση του Μάριο Μόντι μία προσέγγιση που θα βοηθήσει να βρεθεί λύση σε αρκετές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την Ιταλία. Μιλώντα για κρατικέ ενισχύσει, δεν είναι ο τομέα που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα, αλλά είναι, πρέπει να μα απασχολήσει. Ναι, ναι, ναι. Δε, ναι, μα απασχολεί. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερα, αλλά μα απασχολεί. Uh, you, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για την πολιτική ανταγωνισμού και τον τραπεζικό τομέα. Το 2010 ήμουν εισηγητής ε, για την πολιτική ανταγωνισμού και τότε σας είχα θέσει το εξής ερώτημα. Η στήριξη της ρευστότητα για τις περιφερειακές τράπεζες της Ισπανίας και συγκεκριμένα την βοήθεια που είχαν λάβει από την ΕΚΤ γιατί μετά ε, τη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ε, σε κρίση οι τράπεζες, υπήρχε αυτό το, αυτή η φούσκα των ακινήτων και πήραν στήριξη από την ΕΚΤ. Πολύ έξυπνα τότε μου είχατε απαντήσει ότι δεν είναι θέμα για την πολιτική ανταγωνισμό αυτό, γιατί έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική. Ωστόσο, όταν πήραν κρατικές ενισχύσεις οι τράπεζες, αυτό ήταν θέμα πολιτικής ανταγωνισμού. Και έπρεπε να πληρούν διάφορες ε, απαιτήσεις και κριτήρια. Συνεχίστηκε η ιστορία αυτή με τα κάχας, τα πολύ γνωστά, διαβόητα αυτά ε, τα μιευτήρια. Επτά νομίζω κάχας συγχωνεύτηκαν στην Μπάνκια, δημιούργησαν την Μπάνκια. Αν έχουμε 7 τέτοια ταμιευτήρια λοιπόν σε πρόβλημα, είναι αφελέ να θεωρεί κανεί ότι αυτό που προήλθε από τη συγχώνευσή του η μπάνκια δεν θα έχει πρόβλημα. Και έγινε μια too big to fail τράπεζα η μπάνκια ε, που δεν πρέπει να ε, καταρρεύσει να αποτύχει. Θα έπρεπε να τα είχατε δει αυτά τα γεγονότα εδώ και δύο χρόνια. Τα προβλήματα λοιπόν με τα κάχα και με την ε, μπάνκια έχουν να κάνουν, ε, δημιουργούν την ανάγκη διάσωση ε, του ισπανικού τραπεζικού τομέα με ποσό γύρω στα 100 δι. Και ο Ισπανό Πρωθυπουργό αυτό είπε ότι είναι νίκη για το ευρώ. Τι να σα πω εγώ, κλείσουμε λίγο με την παρατήρηση, δεν βλέπω πού είναι η νίκη αυτή. Και πάλι μπορεί να μην αρκέσει αυτό το ποσό. Το ερώτημα μου τώρα είναι λοιπόν, αν δείτε πίσω λίγο. Πώ αντιμετωπίσατε το πρόβλημα των κάχα, των ταπνιστήριων, δηλαδή τη της μπάνκια. Θεωρείτε ότι εφαρμόσατε τη σωστή πολιτική ανταγωνισμού ή μήπως θα έπρεπε να είχατε δραστηριοποιηθεί λίγο πιο ενεργά στον τομέα αυτό για να αποτρέψετε την καταστροφή την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έπιγκ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να με δύο διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι οι επιχειρήσει ε, νομισματική πολιτική τι οποίε αποφασίζει η εκτιστή Φραγκφούρτη. Και πράγματι το έχω πει πολλέ φορέ ότι αυτό είναι νομισματική πολιτική. Άλλη πτυχή εντελώ όμω είναι δημόσια πόροι, δημόσια στήριξη που δίνεται ή πρέπει να δοθεί ε, για την ανδιάθρωση και διάσωση κάποιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μπορεί να είναι τα ταμιευτήρια τα ισπανικά, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό συνασμός, οποιοδήποτε κράτο μέλο. Το πρόβλημα με την Πάνκια, αυτό θέλετε να συζητήσουμε, και επειδή το γνωρίζω καλύτερα γιατί είναι της χώρας μου η τράπεζα αυτή, δεν έχει να κάνει τίποτα με τις ε, πράξεις και τις ε, ΕΚΤ. Ουσιαστικά έχει να κάνει με έγχυση δημόσια στήριξη από την ΕΚΤ που οδηγεί ε, το ότι μπαίνουν στις μετοχές ε, ως ένεση, αν θέλετε, ε, μπαίνει ένα μετοχικό κεφάλαιο, 4,4, υβριδικό συγγνώμη κεφάλαιο, 4,4 δις αν έχω σωστά τον αριθμό στο μυαλό αυτή τη στιγμή και με τη νέα συμφωνία πλαίσιο που ενέκρινε πρόσφατα το Eurogroup, που θα πρέπει βέβαια να γίνει μνημόνιο στην ενόηση επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, και με βάση τις πληροφορίες ε, στα μέσα ενημέρωσης, κατά πάσα πιθανότητα η μπάνκια θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό ε, δημόσιων ενισχύσεων, δημόσια στήριξη. Και όπως έγινε με τα πρώτα 4,4 δις, αυτή η έγχυση δημόσια χρήματος, δημόσιας υποστήριξης θα είναι υπό τον απευθείας, από τον άμεσο έλεγχο της Κομισιόν από τη σκοπιά δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων. Αλλά σας παρακαλώ την νομισματική πολιτική τη ΕΚΤΑ και την έγχυση δημόσιας υποστήριξης ε, μέσω δημοσιοκεφαλαίου ή ε, με οτιδήποτε άλλο ή τις κρατικές εγγύσεις, αυτά να μην τα αναμειγνύουμε το ένα με γιατί είναι διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να στρέψουμε το βλέμμα προς μια, έναν άλλο τομέα του ανταγωνισμού που δεν θίξαμε, συγκεκριμένα στην παροχή τροφίμων. Εκεί είναι ο ανταγωνισμός πολύ σημαντικός ε, γιατί πρέπει οι τιμές τροφίμων να είναι ε, λογικές. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας, ειδικότερα η παραγωγή του γάλατος. Εγώ έχω επανειλημμένως ε, μιλήσει για την ε, περιοχή προέλευση καταγωγής μου, όπου υπάρχουν πολλοί γαλακτοπαραγωγοί και υπάρχουν ε, θέματα ανταγωνισμού. Είναι μικρές οι, ε, οι μονάδες εκεί, οι οποίες έχουν προβλήματα λόγω του ανταγωνισμού από τις μεγαλύτερες εταιρείες, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, υπάρχουν ε, κάποιες ε, προτάσεις για μονάδες παραγωγής, αλλά θα ήθελα να μάθω πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχω πάρα πολλές φορές πει ότι θα ήταν καλό να σταδιακά στην αλυσίδα παραγωγής ε, να επέμβουμε ώστε να υπάρχει ε, μια καλύτερη ρύθμιση των τιμών και να μην υπάρχει σύγκρουση ε, σε επίπεδο ανταγωνισμού. Πραγματικά η Κομισιόν δεν έχει ξεκαθαρίσει όλο αυτό το διάστημα τι προτάσεις έχει για να έχουμε έναν σωστό και αποδεκτό κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. στην έκθεση για τον ε, τομέα των τροφίμων η οποία έγινε με βάση των ε, πολλών δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών ε, σε επίπεδο ανταγωνισμού εφαρμόζοντας τη συνθήκη βλέπουμε όπως το είπα και στην αρχική μου έκθεση, ότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις που ε, αναφέρονται στο άρθρο 100 και 102 της συνθήκης. Είναι αλήθεια ότι μεγάλη πλειοψηφία των παραβάσεων που ανοιχθεύθηκαν και ε, πέστησαν κυρώσεις από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν έχουν να κάνουν με τους ε, κτηνοτρόφους ε, αλλά με τα άλλα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, τους άλλους μεσάζοντες που ασχολούνται με την με, το εμπο... με την ε, προμήθεια του εμπορεύματος του σιταριού, του γάλατος κτλ. Έτσι λοιπόν ε, είναι εκ των υστέρων ε, στην αλυσίδα που υπάρχει το πρόβλημα και όχι στη φάση της κτηνοτροφίας ή της γεωργίας. Αυτό που προκύπτει από αυτή την ανάλυση και αυτό είναι η γνώμη μου γιατί δεν είμαι ειδικό στον τομέα των τροφίμων είναι ότι οι εντάσεις στις τιμές των τροφίμων συχνά βασίζονται σε στοιχεία που δεν σχετίζονται με την μη ύπαρξη ανταγωνισμού ή με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Ε, συνήθως ε, σχετίζονται με θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Τρίτον, αυτό που προκύπτει από την ανάλυση αυτών των αποφάσεων είναι ότι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι εποφελούνται από μία ενεργό και προνοητική στάση των αρχών ως προς τα άλλα στάδια της διατροφικής της αλυσίδας ε, ε, της ε, πώλησης τροφίμων. Από αυτά που κάνουν τα, ε, οι 27 εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ε, βγάζουμε αυτά τα συμπεράσματα. Η Κομισιόν δεν κάνει και πολλά γιατί όλες οι περιπτώσεις ε, παραβίωσης της πολιτικής ανταγωνισμού αντιμετωπίζονται από εθνικές αρχές, εκτός από κάποιες περιπτώσεις συγχωνεύσεων και αντιτράστ δραστηριοτήτων που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό φαίνεται και στην έκθεση που εγκρίθηκε και που ε, συζητάτε τώρα στις συζητήσεις μας. Περισσότερες ε, ε, από τις δραστηριότητες έχουν να κάνουν με αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη ε, στην καθημερινή τους εργασία ως αρχές ρύθμισης του ανταγωνισμού. Λοιπόν, τελείωσε η ομάδα εργασίας, έχουμε άλλους 11 ομίλητες, οπότε τώρα θα σας βάλω σε ομάδες των τριών. Προσπαθήστε να κάνετε απλές ερωτήσεις. Οι τρεις πρώτοι ομιλητές. Ραμόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Αλμούνια. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια ερώτηση. Εθνικοποίηση των τραπεζών καταρχάς. Μέσω της εθνικοποίησης των τραπεζών το εθνικό κράτος γίνεται ο πρώτος μέτοχος της Ιμπέρια, 15% του πακέτου των μετοχών. Η Ισπανία είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου το ε, αεροπορικό δίκτυο ανήκει ε, στο κράτος από την άλλη πλευρά. Όμως είναι ελληματική σε ό,τι αφορά άλλους τομείς της αεροπλοείας. Θα επιθυμούσα λοιπόν να γνωρίζω την άποψη της Επιτροπής. Δεύτερη ερώτηση. Ο πρόεδρος Ραχώη επιμένει σε μία άμεση διάσωση της τράπεζας χωρίς να περάσει από το φρόμπ. Αυτό σημαίνει μία αλλαγή άποψης σε σχέση με τη θέση που υιοθέτησε η ίδια η Επιτροπή. Συγγνώμη κύριε Επίτροπε, τρεις ε, παρεμβάσεις θα ακούσουμε, διαφορετικά χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Παρακαλώ και μετα είπα. με ενδιέφεραν πάρα πολύ τα σχόλια που είχατε να κάνετε. Ε, το θέμα του ανταγωνισμού με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μας βρίσκει σύμφωνους ε, τα όσα έχετε κάνει με, κάνει με το CDS και με τα ε, παράγωγα. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας πείτε κάτι για το κείμενο Μίφιτ και Μιφίτ και τα άρθρα 28, 29 και 30 τα οποία αναφέρονται σε ένα όραμα της Επιτροπής για μια πιο ανταγωνιστική αγορά. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε σε αυτήν την Επιτροπή γιατί αυτή η οι ρήτρε αυτές ε, είναι απαραίτητες για να ρυθμιστούν οι εκαθαρίσεις στην Ευρώπη για να παραμείνουμε ανταγωνιστικές. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντική αυτή η πρόσβαση για την ενιαία αγορά. Ενδεχομένως θα γνωρίζετε ότι η Επιτροπή αυτή υπέβαλε αρκετές τροπολογίες από πλευρά αρκετών μελών για να διαγραφούν αυτές οι ρήτρε πρόσβαση. Συνεπώ θα είναι πάρα πολύ, αναμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλιά σα. Ήβα. Μία ερώτηση σε ό,τι αφορά το μέλλον. για το χρονικό διάστημα 2014-2020, τότε πόσο εσείς και οι υπηρεσίες σας έχετε κινητοποιηθεί έτσι ώστε να μην υιοθετήσουμε πολιτικές που εκτρέπουν τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, αυτά τα προγράμματα που μας απασχολούν στο θέμα της ε, γεωργίας, οι πολιτικές που συζητώνται πολλές φορές ε, κάνουν ε, διαρκείς τις εκτροπές του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μου και τις άμεσες επιδοτήσεις στους γεωργούς, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια περαιτέρω ε, μεταβατική περίοδος. Φτάνουμε στην τέλη 20 χρόνια. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας και πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να κάνουμε πράγματα που συμβάνουν στην εκτροπή αυτή των αγορών. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τις ερωτήσεις, κύριε Τρεμός, πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να προδικάσω, να προκαταλάβω κάτι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία επίσημη απόφαση, ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε κοινοποίηση. ούτε για το μέλλον των ε, βιομηχανικών συμμετοχών της Μπάνκια στο σχέδιο μιας αναδιάρθρωσης. Θα το αποφασίσουμε, θα δώσουμε την άποψή μας, ούτε έχει υπάρξει, επαναλαμβάνω, κοινοποίηση ότι οι Ισπανικές αρχές ενδέχεται να ξαναθέσουν θέμα ιδιωτικοποίησης ή αλλαγής ε, σε σχέση με τον εθνικό αερολιμένο διαβάζουμε εφημερίδες και εσείς και εγώ στις χώρες μου και τα διαβάζουμε αυτά. Έχουμε περιπτώσεις ανδιάρθρωσης λιμένων, Έχουμε περιφερειακά ε, που γίνονται τοπικά. Έχουμε κάποιες επιδοτήσεις ε, συγκεκριμένων ε, που, εταιρίων που χρησιμοποιούν τα τοπικά ή περιφερειακά αυτά αεροδρόμια. Σε κάποια έχουμε κάποιες προσφυγές, σε κάποια έχουν ανοίξει. Δεν έχω να πω τίποτα για την απευθείας άμεση διάσωση. Είναι μια ε, επιλογή την έχει αναφέρει και από τη κυβέρνηση το έχω διαβάσει και στα μέσα ενημέρωσης ε, από το Μεξικό μέχρι και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν ε, μεταφέρονται σωστά όλα αυτά τα οποία γράφονται. Υπήρξε σχέδιο διάσωσης μια σειρά τραπεζών που συμφωνήθηκε την πρώτη εβδομάδα στο Eurogroup με βάση τις αναλύσεις που έχουμε μέχρι τώρα με την νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ίσως υπάρξει όμως τροποποίηση κάποια στιγμή αυτής της νομοθεσίας. Αλλά προς το παρόν μιλάμε για συνθήκη μηχανισμό, διακυβερνητικό μηχανισμό σταθεροποίησης. Ε, δεν έχει δικαίωμα πρωτοβουλία η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για το MIFID MIFID, ο κύριο Παδάρη κάνει τη σχετική ερώτηση. Εγώ δεν είμαι αρμόδιο για τι κρατικέ ενίσχυσει στο γεωργικό τομέα. Γεωργία και Αλία ε, εξαιρούνται από το γενικό κανόνα. Οι συνάδελφοι τη Γεωργίας και συγκεκριμένα ο Επίτροπο Τσόλο ε, για τη Γεωργία και ο Επίτροπο Δαμανάκη για την Αλία είναι οι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Μίφιντ, μίφιρ. Δεν μπορώ να σα απαντήσω λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνω είναι αρμοδιότητα άλλων συναδέλφων επιτρόπων. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, δική μου θέση και άποψη για την ανοιχτή ελεύθερη πρόσβαση σε δραστηριότητε συμψηφισμού, clearing ε, ή σε κάποιους ε, κεντρικούς ομολόγους. Εγώ στηρίζω απόλυτα την πρόταση της Κομισιόν. Γνωρίζω ότι τώρα δική σας είναι η ευθύνη, από δικη σας ειναι η ευθυνη απο με το Συμβούλιο να συζητήσετε και να νομοθετήσετε στη δική μας πρόταση. Σεβόμαστε πλήρως την αρχή της μη διακριτικής πρόσβασης. Γενικώ. Και σε ό,τι αφορά τα license benchmarks. Αυτές ήταν οι αρχές και γι' αυτό είχαμε και μια αρνητική απόφαση για την Deutsche Börse Neise και μπορείτε να τη μελετήσετε για να λάβετε και τις κερδικές αποφάσεις. Εμείς ε, βασιζόμαστε σε αυτή την αρχή. από την αρχή της ελεύθερης μη διακριτικής πρόσβασης. Δεν έχω όμως εγώ αρμοδιότητα να επηρεάσω αυτό το οποία θα συζητήσει και θα τα αποφασίσετε εδώ. Ευχαριστώ. Οι επόμενοι τρεις... Ε, δεύτερη κυρία Κράτσα. Ε, Ευχαριστώ, ε, Επίτροπε Αλμούνια. Βλέπουμε ότι πολλοί ε, πολίτες σέβονται την εργασία σας, ε, κατανοούν ότι η αρχή της ανταγωνιστικότητας είναι ο καλύτερος φίλος του ανταγωνισμού και ότι οι επιχορηγήσεις και οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι προς συμφέρον τους. Επίσης, δεν θέλουν οι ε, είτε συμφωνούν είτε όχι με την διάσωση των τραπεζών, δεν θέλουν οι τράπεζες ε, να πτωχεύουν. Ε, καταλαβαίνουν την ανάγκη. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια εθνική, ας πούμε, μικρή εταιρεία στον τομέα της αεροπλοίας, για παράδειγμα, που είναι στρατηγική για τη χώρα, είναι η μοναδική ας πούμε εταιρεία που εκτελεί ένα συγκεκριμένο ε, ρόλο. Ε, λαμβάνει κρατικές ενισχύσεις, αλλά όταν βλέπουν ότι η απάντηση σχετικά με τις δραστηριότητες, δυνατότητες αναδιάρθρωσης παίρνει πολύ χρόνο, δεν κατανοούν γιατί αυτό συμβαίνει. Κυρία Ροδικράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Αφενός θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι αποτιμήσεις που έχετε κάνει, εξολογήσεις για τη λειτουργία των επιτροπών, ανεξάρτητων επιτροπών αρχών ανταγωνισμού στις διάφορες χώρες. Ε, υπάρχει πράγματι αυτή η ανεξαρτησία. Ε, Ποιε είναι οι χώρες και πού οφείλεται στο ότι υπάρχουν στρεβλώσεις σε μερικές χώρες από παρεμβάσεις κρατικές. Ε, δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω στις χώρες με προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής παρατηρείται η δυσκολία στη χώρα, παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα, το βλέπουμε, ότι υπάρχει δυσκολία να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, διότι συνεπάγεται μεταρρυθμίσεις, αλλαγές που ε, σε, στην περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι δύσκολο να απορροφηθούν και από την αγορά και από την κοινωνία. Ε, βλέπετε να υπάρχει πρόοδος, χρειάζονται συμπληρωματικές ε, παρεμβάσεις από την πλευρά σας στις περιπτώσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω, να σας ε, συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας θέσω και κάποιες ερωτήσεις. Ε, έτσι έχω ρίξει μια ματιά στην έκθεση που μας υποβάλλατε και στην ανάλυση των μικρών αξιολόγησης. Λέτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ε, κάποιων δραστηριοτήτων ή ενεργειών κατά του ανταγωνισμού. 2009 λέμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Μιλάμε για ένα σύστημα υποχρεωτικής ε, εναλλαγής, περιτροπής. Δεν ε, πιστεύετε ότι πρέπει να δούμε και το ρυθμιστικό σκέλος, δηλαδή δεν θα ήταν καλύτερα το πρόβλημα του ανταγωνισμού να το δούμε στο πλαίσιο του δικαίου ανταγωνισμού να ξεκινήσει μια τομεακή ανάλυση, να δούμε υπήρξαν παραβιάσεις και αν ναι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Πρώτο, δεύτερο ερώτημα, αεροπορία. Υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ αερομεταφορέων. Υπάρχει μια περίπτωση, τη γνωρίζω πολύ καλά, με την Brussels Airlines και την TAP με πτήσεις ε, Πόρτο Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει και σχετική έρευνα. Τι γίνεται λοιπόν ε, με το σκηνούς κωδικούς πτήσεων σε αυτό το δρομολόγιο. Ευχαριστώ. Well, regarding the, the first question... Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, Understood exactly. δεν κατάλαβα ακριβώς αν αναφράσασταν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση ανταγωνισμού. Εάν ναι, μπορώ να απαντήσω. Λέει ναι, βλέπω. Νεύει, νεύει καταφατικά. Ωραία, άρα μπορείτε να μου το διευκρινίσετε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δύο ερωτήματα που αφορούν τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Δεν έχουμε νομική ε, εξουσία και αρμοδιότητα για να τροποποιήσουμε ή να μετασχηματίσουμε τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες υποχρεούνται να επιβάλλουν το άρθρο 101 και 102 της συνθήκης. Διατηρούμε μαζί τους επικοδομητική και αποδοτική συνεργασία και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. και στο τέλος ε, της νομικής διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν ε, μια συγκεκριμένη εθνική αρχή ανταγωνισμού εφαρμόζει σωστά ή όχι τη συνθήκη. Υπάρχουν βέβαια κάποιε απόψει. Κάποιε εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού έχουν καλύτερη χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προπολογισμού, άλλε δεν είναι τόσο ανεξάρτητε απέναντι στις εθνικές αρχές, στην κυβέρνηση δηλαδή. Αλλά για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η έκβαση, είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή εφαρμόζει σωστά τους κοινούς κανόνες που πρέπει, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε η εκάστοτε Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού. Και το βλέπουμε αυτό και στην κατανομή των υποθέσεων. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ επικοδομητική συνεργασία με όλες τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις Διερωτώ με μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις συστάσεις χώρα ε, στο πλαίσιο δηλαδή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ανταγωνισμού εργάζονται. Φέτος, νομίζω ότι οι συστάσεις τουλάχιστον σε μία περίπτωση αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού. Είχαμε λοιπόν συστάσεις προς μία χώρα και πίσω στο πλαίσιο των προγραμμάτων για Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, εκεί εισαγάγαμε κάποια σχόλια και κάποιες σκέψεις για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά δεν απατώμε και στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε, αυτή τη μόχλευση ε, για να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργούν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τους οίκους αξιολόγησης, Είμαι βέβαιος ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να βελτιωθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που εργάζονται αυτοί οι Ε, Είμαι πεπισμένος προς αυτό. Μέχρι στιγμής όμως νομίζω ότι το καλύτερο μέσο για τη βελτίωση των ανταγωνιστικών αυτών πτυχών των οίκων αξιολόγηση είναι ο κανονισμός η ρύθμιση. Περισσότερο ρύθμιση και όχι τόσο η πιθανή χρήση μέσω, αντιμονοπολιακών μέσων και εργαλείων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει ούτε μία καταγγελία γι' αυτό. Ούτε έχουμε βρει επιχειρήματα για να ξεκινήσουμε αυτά επάγγελτα με βάση το άρθρο 101 ή το άρθρο 102 της συνθήκης κάποια έρευνα όπως γνωρίζετε βέβαια, γιατί το απεξεργάζεται αυτό το θέμα το Κοινοβούλιο, η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται ενεργά ε, στο θέμα ε, των ε, ρυθμίσεων για τους οίκους αξιολόγησης. Έχουμε τρία θέματα, rotation, το είπατε και άλλα. Αυτά τα περιλαμβάνουμε στις ρυθμιστικές προτάσεις, όπως είπα στον αριθμό, ό,τι αφορά την αεροπορία. Πράγματι, ε, μελετούμε κάποιες συμφωνίες ε, κοινή χρήση κωδικών, code share, ε, κάποιων αεροπορικών εταιρείων σε κάποια δρομολόγια, ένα από τα οποία είναι αυτό το οποίο αναφέρατε με συμφωνία TAP Brussels Airlines. Πρέπει να σας πω ότι εάν είναι καλές πληροφορίες που έχω, το 70% των εσωτερικών δρομολογίων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται από μία μόνο εταιρεία. The question from the competition point of view... Δυστυχώς δεν είναι σαφές αν λέει 17 ή 70. Ο κύριος Αλμούνια. Λοιπόν, αν υπάρχουν καταχρήσεις θα το δούμε, αν υπάρχει κατάχρηση δεσπόσιας θέσης, αλλά θα πρέπει να δούμε και αν υπάρχει αν υπάρχουν φραγμοί ε, στην πρόσβαση και έρχομαι, πάλι στην ερώτηση Χέλμαρκ για την πρόσβαση και για τους φραγμούς. Σε πολλά δρομολόγια δεν, υπάρχει, δεν είναι θέμα το αν υπάρχει ε, ε, πρόβλημα στην πρόσβαση για να ασχοληθεί κάποιο με αυτό το δρομολόγιο, αλλά ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Ευχαριστώ. Just what, what I'm saying is that's what, what the constituents say. Αυτό που λέω είναι, αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, ότι όταν παρακολουθούν ε, τα δισεκατομμύρια που δίνονται στις τράπεζες, γνωρίζοντας ότι αυτά πάνε από την τσέπη τους, θέλουν να βοηθήσουν ε, μια στρατηγική όμως ε, αεροπορική εταιρεία ε, θέλουν να το κάνουν. Υπάρχουν ε, λοιπόν στιγμές που χρειάζεται αναδιάρθρωση και θα το κάνουν. Αυτό λένε. Ε, εργαζόμαστε στο θέμα της, ε, των γραμμών της Μάλτας και τώρα θα πλησιάσουμε στο τέλος. Σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις είχαμε όλα τα εργαλεία στα χέρια μας. Εάν τα άλλα μέρη, αυτή τη στιγμή μιλάω για τις εθνικές αρχές ε, δεν μας δίνουν τις ε, πληροφορίες που θέλουν ή αν ε, το σχέδιο αναρδιάρθρωσης που τους δι, μας δίνουν δεν συμφωνεί με τους κανόνες ανταγωνισμού πρέπει να, έχουμε, να ζητήσουμε ένα σχέδιο, επιπλέον πληροφορίες έτσι ώστε στο τέλος να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Το θέμα με τις τράπεζες, το ξέρουμε. Έχουμε πρόβλημα, ίσως τους περισσότερους από τους άλλους οικονομικούς τομείς μπορεί να φανταζόμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτόν τον τομέα και χωρίς αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Στην περίπτωση του οικονομικού συστήματος παίζει τόσο σημαντικό ε, ρόλο που δεν μπορούμε να ζήσουμε, να αναπτυχθούμε, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας χωρίς ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που δεν μπορεί ε, ε, που να μπορεί να χρηματοδοτήσει να υποστηρίξει. Γι' αυτό λοιπόν στην χρηματοπιστωτική κρίση κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες προσπαθώντας με υποστήριξη από το κοινό, με μοίρασμα των, του, του άχθους όσο γίνεται. Τέλος, οι τελευταίες τρεις ε, ερωτήσεις Βέρνερ Λάγκεν, ε, Μαρτά και Ρομπέρτα Καλτιέρη. Βέρνερ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω μία επερώτηση σε σχέση με αυτά που αναφέρατε για τη συγκεντρώση στα καρτέλ. Αν τα, αν τα κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν είναι τα καρτέλ στα τρόφιμα, αλλά ε, στην ε, πρόθεση των δεν ξέρω τι γίνεται με την κορδοσκοπία πρώτων υλών. Η δεύτερη ερώτησή μου, μιλήσατε για την ε, Bayerische Landesbank. Υπάρχει περίπτωση ε, η Dexia, η Societe Generale, που μέσα σε 24 ε, ώρες δώσατε άδεια για αυτή την συγχώνευση. Υπάρχουν τώρα νέες ε, περιπτώσεις ε, όπου η διάρκεια της διαδικασίας ε, επαλήθευσης είναι μεγάλη. Έχουμε από την Ιρλανδία τη Μερκλέρ, η οποία έχει διαδικασίες πάνω από τέσσερα χρόνια για τη Ryanair, και δεν μπορεί να πετάξει σε διάφορα ε, αεροδρόμια και λέει ότι δεν θα φτάσουν ε, αυτές οι διαδικασίες ε, στο τέλος. Μπορείτε να μιλήσετε και να μας πείτε κάτι σε σχέση με αυτές τις αιτιάσεις, γιατί διαρκούν τόσο πολύ οι διαδικασίες. Μάρτα. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτρεπε, μιλήσατε για ένα καλό προηγούμενο σε σχέση με τις έξι τράπεζες που είναι υπό αναδιάρθρωση. Είναι μόνο αυτά τα κακανέα που θα πάρουμε από... για τις τράπεζες, γιατί τα stress tests δεν βλήκανε από ό,τι φαίνεται τις προβληματικές τράπεζες. Όταν έχουμε χρήματα που δίνονται σε τράπεζες χωρίς να γίνεται διερεύνηση των λόγων που ε, τις οδήγησαν σε αυτό, αυτή την ε, δινή θέση δεν φαίνεται πολύ δίκαιο από άποψη ανταγωνισμού. Μάλλον ε, υπήρχε ανευθυνότητα στη διαχείριση των τραπεζών. Ε, τι γίνεται όταν το διαπιστώσουμε αυτό, θα πρέπει να διασώζονται οι τράπεζες αυτές, ε, καθώς αυτό ε, επιδεινώνει το χρέος ε, και το ποσοστό ελλείμματος της χώρας. Άλλο ερώτημα. Πριν ε, γίνετε επίτροπο ανταγωνισμού, ήσασταν επίτροπο νομισματικών και οικονομικών υποθέσεων. Η κρίση τώρα είναι αποτέλεσμα διαφόρων ε, παραγόντων, όπως και το μέσα σε αυτούς ε, και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κομισιόν. Αποδέχεται η Κομισιόν τις ευθύνες γι' αυτό. Έχετε βρει κάποια στοιχεία, κάποιου κανονισμού που να είναι λανθασμένοι και τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτούς. Ρομπέρτα. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα, μόνο ότι θα ήθελα να το δω από γενική άποψη. Η έρευνα που ξεκίνησε η Επιτροπή για την Προαναγγελθή Θήσα αγορά τη σύνοξου Ματσάι Σπετσάλι από την, ε, τον όμιλο Τίσεν. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία, δεν θα ήθελα να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Είναι επίσης ε, ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία αφορά έναν από τους μεγαλύτερους ε, παραγωγούς χάλιβα στον κόσμο και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Η ερώτησή μου αφορά τη συγκεκριμένη βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο υφίσταται η ισορροπία μεταξύ των δύο αρχών του άρθρου 101 τη συνθήκης. Η βιομηχανία αυτή είναι μια βιομηχανία όπου ο ανταγωνισμός προέρχεται από το εξωτερικό. Το 50% της παραγωγής είναι στην Κίνα. Και διαδικασίες σαν και αυτή θα μπορούσαν να, να θεωρηθούν διαδικασίες εξυγίανσης του προπολογισμού όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα που διατρέχει σοβαρό κίνδυνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 101 που απαγορεύει τις συμφωνίες που εκτρέπουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και του δεύτερου που λέει ότι δεν εφαρμόζεται αυτή η απαγόρευση σε όλες τις συμφωνίες οι οποίες συμβάνουν στη βελτίωση της παραγωγής ή συμβάνουν στη τεχνική πρόοδο. Yes. Ναι, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία. Ε, α, στα ισπανικά θα απαντήσω. Ε, Παντώ λοιπόν στον κύριο Λάγκεν. Η διάρκεια ε, για περίπτωση κρατικών ενισχύσεων αλλά και αντιτράστα, αλλά εσείς μιλήσατε για κρατική ενίσχυση. Εδώ αυτό εξαρτάται από τη μία από την πολυπλοκότητα τη εκάστοτε υπόθεσης που θα πρέπει να αναλύσουμε και το είδο τη ενίσχυση που δόθηκε ή θέλει να δώσει το κράτος μέλος. Εξαρτάται επίσης από την άλλη πλευρά και από τη συνεργασία που έχουμε με το και ο κράτος μέλος που είναι και ο μόνος ε, δια, ε, συνομιλητής μας όταν ανοίγει η υπόθεση. Αν προχωρήσουν οι έρευνες, εκεί ναι μπορούμε να απευθυνθούμε και σε άλλους ενδιαφερομένους φορείς, αλλά αρχικά μόνο στο κράτος μέλος. Αυτό είναι ο συνομιλητής μας, μόνο. Και έπειτα υπάρχουν φορέ, πολλές φορές ε, ε, δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη έχουμε κρατικές ενισχύσεις που είναι απόρρια μιας απόφασης του δικαστηρίου που μας υποχρεώνει να ξανανοίξουμε την υπόθεση όπως με τα γερμανικά ταχυδρομεία, Deutsche Post. Αλλά τις προάλλες σε μια συνεδρίαση εδώ, σε ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκα σε αλλαγή της διαδικασίας που θέλω εγώ να θεσπίσω στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού ε, του καθεστώτος ε, κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή, να μπορούμε άμεσα και απευθείας να απευθυνόμαστε σε κάποιον που θα μπορεί να μας δίνει πληροφορίες. Αν το οικείο κράτος μέλος δεν μας αποστέλει αυτές τις πληροφορίες. Και ένας εκπρόσωπος ε, ενός κρατηδίου, ε, όχι του δικού σας κύριε Λάγκεν, αλλά τόσο πάνω ενός ομοσπονδιακού κρατηδίου της Γερμανίας μου είπε ότι είμαι κατά, εντελώς κατά. Ο μόνος που πρέπει να δίνει πληροφορίες πρέπει να είναι το οικείο κράτος μέλος. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο για να σεβαστούμε αυτή τη σχέση συνομιλητή που έχουμε με το κράτος μέλος που έδωσε ή ε, θέλει να δώσει την κρατική ενίσχυση, αλλά σίγουρα πρέπει ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και να επιταχύνουμε και την επίλυση των ε, υποθέσεων. Στην προκειμένη τώρα περίπτωση που μου αναφέρατε, εμείς κάναμε κάποια βήματα προς τα εμπρός, κάποια πρόοδο ε, έχουμε ήδη επιτελέσει, είναι μακρά η διαδικασία και έχουν ξεκινήσει ήδη Επόμενη παρέμβαση. Τα stress test δεν είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου Ανταγωνισμού, ούτε καν τη Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικοί επόπτε, ε, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είναι αρμόδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμετείχε σε κάποια ε, τεστ αντοχή αυτή, με υποθέσει, δηλαδή παρέχοντα υποθέσει εργασία, αλλά δεν είχε άμεση συμμετοχή στη διεξαγωγή ενό stress test που επαναλαμβάνω οι επόπτε είναι που έχουν την αρμοδιότητα. Ότι χρειάζεται βελτίωση Συμφωνούμε όλοι, είδαμε ότι κατά το παρελθόν σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα τα πράγματα και στη μεθοδολογία και στα αποτελέσματα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να αναλύουμε την τράπεζα, την εκάστοτε τράπεζα σε κάθε περίπτωση κρατική ενίσχυση, γιατί κάνει κάθε τράπεζα. Αυτό δεν είναι δική μα αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά εμεί αυτό που μελετάμε είναι γιατί ζητάει χρήματα. Θα πάρει κάποια χρήματα. Πρέπει να έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που να είναι βιώσιμο. Πρέπει να πάψουν επιζήμιες πρακτικές για τη φερεγγιότητα κτλ. Επιχρεώνει να γίνουν επενδύσεις, ε, να αλλάξουν ε, μέθοδοι διαχείρισης, ε, να αλλάξει χρηματοδότηση κτλ. λοιπά. Αυτά περιλαμβάνονται στην συζήτηση του επιχειρηματικού μοντέλου και έτσι μπαίνουμε και στην ουσία, μπαίνουμε στο βάθος. Βέβαια, εκτός αν η πρόταση του σχεδίου αναδιάτρωσης που διατυπώνει το ε, κράτος μας που δίνει δηλαδή την ενίσχυση, αν αυτά περιλαμβάνει, δεν μπορούμε με δική μας απόφαση να πούμε τίποτα στους, ε, στη διοίκηση, στους μάνατζερ. Σίγουρα καλό θα ήταν να αντικατασταθούν οι κακοί ε, διαχείριστες από καλούς, αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, παρότι θα ωφελούμε θα όλοι από αυτό. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε μονομερός να αλλάζουμε τους μάνατζερ εμείς σε κάποια εταιρεία ή σε οποιοδήποτε οργανισμό. Επίσης, με ρωτήσατε για το νομικό πλαίσιο της ΟΝΕ. Μάλλον στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνεται αυτό το ερώτημα, γιατί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ορίζουν αυτό το πλαίσιο και όχι Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κουαλτιέρη με ρωτήσατε για μια υπόθεση την οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή και είναι στη φάση 2, αν δεν με πατάει η μνήμη μου το σχέδιο εξαγοράς αυτών των εργοστασίων ανοξίδωτου άνθρακα της Τίσεν στο Τιμπουκτού. Αυτά τα συζητούμε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, λίγα λεπτά απομένουν μόνο. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να επεκταθείτε λίγο σε ένα-δυο πράγματα που Ο Βέρνερ θέλει κάτι να πει. Δεν απαντήσαν σε ερωτήσεις σας. Είχα θέσει και άλλες δύο ερωτήσεις. Δεν ξέρω, είτε δεν μπορούσατε, δεν ήθελα να τις ο Επιτροπός. Η μία αφορούσε το Embayer Islandes Bank, μια τράπεζα του κρατηδίου της Βαβαρίας ε, και κάμπεσέ και τα λοιπά. Και το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τις ε, διαδικασίες κατά των καρτέλ στην ε, βιομηχανία τροφίμων. Συγγνώμη, το είχα ξεχάσει αυτό. Όταν ξεκίνησα την κουβέντα μαζί σας ήταν το πρώτο πράγμα αυτό που μου ήρθε στο μυαλό. Και βυσί. Η τράπεζα εφαρμόζει το πρόγραμμα εξυγείας σύμφωνα με την απόφαση που και το 2009. Και όπως σας είπα και προηγουμένως δεν αναφέρθηκα στην KBC αλλά μεταξύ των άλλων στην KBC διαπραγματεύτηκαμε μία αλλαγή σε ορισμένες επενδύσεις. Σε γενικές γραμμές όμως το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης εφαρμόζεται και είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι και ελπίζω ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα μέχρι το, το τέλος. Η LB δεν μπόρεσε μέσω των Ομοσπονδιακών Αρχών, των Βαβαρικών Αρχών, να καταλήξει σε μία συμφωνία σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Το πλησιάσαμε, πλησιάσαμε πολύ αυτό το σημείο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν ορισμένες αλλαγές. Πραγματικά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης του σχεδίου αδιάθρωσης με διάφορους συνομιλητέ κυρίως από την ε, βαβαρική πλευρά και η Επιτροπή και οι Ομοσπονδιακές Αρχές στη Γερμανία εργάζονται σκληρά για να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Και τα καρτέλ, τα καρτέλ στον τομέα των ειδών διατροφής δεν θυμάμαι τι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι στην έκθεση ότι, όπως ανέφερα προηγουμένως, ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καρτέλ που αποφασίστηκαν από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την περίπτωση ενός καρτέλ ευρωπαϊκών διαστάσεων στον τομέα των ειδών διατροφής. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάπως διεξοδικότερα αυτό το θέμα σε σχέση με τις αρχές ανταγωνισμού. Είπατε ότι η Επιτροπή ενδεχομένως θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιήσει συστάσεις εξατομικευμένες για την κάθε χώρα, έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη εξειδράσεις. Τώρα, σε απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα, Είπατε ότι δεν μπορούσατε να ελέγξετε τα όσα κάναμε στην διαδικασία, στην νομοθεσία συναπόφαση. Πράγμα που είναι αλήθεια. Και πραγματικά με ενδιαφέρει η αλληλεπίδραση που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ τη συνθήκη, κοιτάξτε το άρθρο 19, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικές πολιτικέ ω στόχο στα πλαίσια μια ανοιχτή οικονομία τη αγορά. Έχουμε μία σειρά από συστάσεις τώρα ε, που λένε ότι ο τομέας των υπηρεσιών θα πρέπει να ανοίξει και η πρόκληση είναι κατά, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτή ε, πρόσβαση. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οικονομική διακυβέρνηση της συνθήκες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Πιστεύω και το συζητήσαμε το θέμα αυτό και σε διάφορες περιπτώσεις Συμφωνώ απόλυτα και ξέρετε πόσο απόλυτα συμφωνώ με το αίτημα αυτό για μια ανοιχτή οικονομία, ανοιχτή πρόσβαση υπηρεσίε και στον ανταγωνισμό. Όσο είναι δυνατόν, όσο περισσότερο γίνεται μεταξύ των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και μέσων. Αυτό που δεν μπορώ να σας ε, υποσχεθώ είναι ότι θα καταφέρω να πείσω και του 27 υπουργού Οικονομικών και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν κατά 100% τις προτάσεις της Επιτροπής. Γιατί οι προτάσεις της Επιτροπής από αυτή την άποψη όπως αναφέρθηκαν από το μέρο, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το ΜΥΦΙΤ, πλήρω είναι πλήρως συμμορφωνές με αυτό τον στόχο και αναφέρονται στο, σε όλο το τομέα των υπηρεσιών, όχι μόνο το τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ζήταμε από τις χώρες μέλη να είναι πολύ πιο φιλόδοξες όταν εφαρμόζουν την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Αυτό είναι ένας τομέας που θα μας βοηθήσει περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα να κατακτήσουμε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι στον τομέα των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως είπα στην αρχική μου παρουσίαση, όχι μόνο μέσω του ελέγχου των συγχωνεύσεων, αλλά και σε ορισμένες σημαντικές περιπτώσεις αντιτράστα. Μερικές από αυτές είναι ε, γνωστές, σε άλλες ε, αναφέρθηκα ε, ακροθυγός. Ε, είπα όμως ότι είναι περιπτώσεις που μας απασχολούν και θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο μου καθήκον είναι να διαβάσω το χρονοδιάγραμμα. Καταρχάς, Έχουμε ε, στις 20 Ιανουαρίου, ε, στις 20 Νοεμβρίου θα υποβληθεί η έκθεση για την, ε, τον ανταγωνισμό. Περιμένουμε το σχέδιο ε, έκθεσης 17 Ιουλίου. Αυτό θα συζητηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε το ετήσιο εργαστήριο της τις πολιτικές ανταγωνισμού στις 18 Σεπτεμβρίου. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν στις 20 Σεπτεμβρίου και ε, μετά θα εξεταστούν από την Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί στην ε, ΕΚΟΝ στις 20 Ιανουαρίου και ε, μετά θα συζητηθεί στις 13 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι η έκθεση πρωτοβουλία καλύπτει διάφορα στοιχεία ανταγωνισμού. Δεν αποτελεί μόνο απάντηση στη δική σας έκθεση περί ανταγωνισμού. Έχετε πάρα πολλά να πείτε για το θέμα του ανταγωνισμού. Τι είναι η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Όπως πάντα μας διαθέσατε το χρόνο σας και μας δώσατε και πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ένα-δύο λεπτά για να περάσουμε στην ψηφοφορία. Για δέστε τις κάρτες σας. Είναι όλα εντάξει. Okay, um, if you could plug your cards in and uh, do a test vote so we know everything. Λοιπόν, βάλτε τις κάρτες σας να κάνουμε μία δοκιμή, να δούμε αν όλα λειτουργούν. Για πατήστε τα κουμπιά σας παρακαλώ. See how many people have voted on this one. Okay, so far I think we've got 40 cards planned. Έχουν μπει 40 κάρτες, ψήφισαν 41 κάρτες. 33 ψήφισαν, 34, 35, 36, 37, 38. Τι φταίει το σύστημα, τα δω, τα δάχτυλά σας, 42. Τρεις δεν ψήφισαν, δύο δεν ψήφισαν, ένας δεν ψήφισε. Εντάξει. Ωραία, ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, ενημερώθηκα ότι υπάρχουν 41 ευτυχισμένα άτομα εδώ. Έχουμε δύο επιπλέον προφορικές πρωτοβουλίες. Να δώσω λόγο στον κύριο Κλίν. Γιατί δεν έχουμε αντίγραφα. With that proviso, are we... Εντάξει, έτοιμοι είμαστε. Συμβιβασμός A. Yeah, this is the regulation. Yeah? Okay. Um, compromise A. All those in favor. Συμβιβασμός Α. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε. Uh, that is carried 35 in... Εγκρίνεται 35 υπέρ, 8 κατά. Συμβασμός σε β, σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό C. Γάμα, δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα σε μια προφορική τροπολογία από το Άλτε, τους φιλελεύθερους, αλλά θα τη δείτε στο έγγραφο κάτω από τον συμβιβασμό C. Όχι. Όχι, είναι προσθήκη. Ε, για προσθήκη των λέξεων or mechanistically ή μηχανιστικά στο 5α ε, συμβιβασμό C που μόλις ψηφίσαμε. Σωστά. Ποιοι είναι υπέρ της προσθήκης αυτών των λέξεων or mechanistically. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στο συμβασμό D, δέλτα, υπέρ. Να περιμένετε. I'm just Να βρούμε λίγο τη σειρά. Θα ψηφίσουμε πρώτα το συμβασμό. Χωρίς την τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα για προσθήκη των λέξεων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε διάφορα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στο συμβιβασμό ε, που είναι απλώς υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 2 6 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 υπέρ 18 κατά. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η προφορική τροπολογία στο συμβασμό Ε που είναι μια-δυο παράγραφοι που προστίθενται. Όσοι είναι υπέρ της ε, προφορικής τροπολογίας, να το πούν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στον G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. H, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα πάμε στην ε, τροπολογία 308. Έχουμε και την προφορική τροπολογία μαζί. Όχι, ωραία. Πρώτα η τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ της, της βασικής, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ποιοι είναι υπέρ των προφορικών αλλαγών. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Μαζί με την προφορική τροπολογία. Τροπολογία 31. Θα να αποσύρω την 31. Ο εισηγητής απέστειλε την 31. Καταπίπτουν οι άλλες δύο, άρα πάμε στο συμβιβασμό J. Που έχει και μια προφορική τροπολογία. Στο πρώτο μέρος. Θες να εξηγήσεις. Προτείνω να προσθέσουμε κάτω από το 2α for unsolicited credit ratings κτλ. κτλ. Πριν από... που δεν έχουν ζητηθεί για ε, αξιολογήσεις που δεν έχουν ζητηθεί. Υπάρχει κανείς που αντιτίθεται. Αφού ψηφίσουμε το πρώτο μέρος, προτείνω να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Όπως κάναμε και πριν, για το πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η αλλαγή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 273 που είναι διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός K, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται προφορική τροπολογία που έχετε από το άλτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,98, όχι. Όχι. 2,98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το έλκ ήταν υπέρ. Ναι, άρα εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο 2,99 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτή τη φορά διόγκο. 331 υπέρ κατά αποχές Ξανά απορρίπτεται, Χριστέ μου. 3.32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3.34 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 3.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.42 με την προφορική τροπολογία, η βασική πρώτα τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αλλαγή της τυποποίησης σε εναρμόνιση. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της αλλαγής. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 344. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 345. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 346. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στο 367 υπέρ 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία από την ΚΟΕ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε τώρα στο συμβιβασμό π. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Δεύτερο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 381. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μόνο το μέρος το δεύτερο του 381. Πού είμαι. Είμαι ακόμη εδώ. 38 corresponding 38 εγκρίνεται. Και μετά 381 εγκρίνεται και τώρα είμαστε στο συμβασμό Q. Ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 382 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. 383 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 384 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 385 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός R σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 407 στην αρχή της επόμενης σελίδας. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 408 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός τι. Με προφορική τροπολογία. Βολφ, θέλεις να εξηγήσεις την προφολογία σου. Θα ήθελα να προσθέσω τις ακόλουθες λέξεις οι αξιολογίες πιστοληπτικής ικανότητας και προβλέψεις θα πρέπει, θα προσθέτονται επίσης. Το also, δηλαδή το επίσης σε αριθμούς και τα λοιπά. Όχι αποκλειστικά λοιπόν exclusively, αλλά also επίσης. Ε, πρώτον, θα πάρω το πρώτο μέρος και μετά θα ψηφίσουμε για το also. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και για το όλσο τώρα το επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο συμβιβασμό U. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός V. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβασμός W. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 405, ε, 425. Υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβασμός 6. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβασμός Y. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 που, είναι, που συνάδει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 60 περ κατά αποχές να ελέγξουμε την 60 voted? Votes closed. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 23 υπέρ, 22 κατά. Η τροπολογία 60. Τροπολογία 2 υπέρ όχι καταπίπτει 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός AA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας, έκανα λάθος, εγκρίνεται 27 υπέρ, 17 κατά. Μάλλον λάθος, διάβασα τη μία ομάδα. Αιτιολογική σκέψη, τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Α, είχε καταπεί πέσει και την απορρίψαμε. Εκατόν δεκαπέντε. Oh, it Καταπίπτει. Όλες καταπίπτουν. Ωραία. Όλες καταπίπτουν αν εγκριθεί η 4. Έτσι λέει, ε, το οποίο δεν γίνεται γιατί έχει εγκριθεί ο συμπασμός R. Αλλά δεν ξέρω. Ο εισηγητής λέει ότι καταπίπτουν. Άρα 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Έχει καταπέσει 122 καταπίπτει 123. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 καταπίπτει τροπολογία 6 μόνη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προφορική τροπολογία για διαγραφή κάποιων λέξεων από τον εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 127 δεν εγκρίθηκε άρα πρέπει να ψηφίσουμε και τις 128 κτλ. Πάμε πίσω τότε πάλι. Έχετε δίκιο στην 128. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 130 καταπίπτει, 131 καταπίπτει. Θέλετε να ελέγξουμε την 129. Να ελέγχουμε την 129. Την ψηφίζουμε την 129. Yeah, Έχουμε άλλες τέσσερις. Τρεις. Θα κλείσω την ψηφοφορία. Τελευταία ευκαιρία να πατήσετε το κουμπί σας. Εγκρίνεται 26 υπέρ 18 κατά. Αυτές πέφτουν 133, την ψηφίσαμε. Εκτός σειράς, 134. Καταπίπτει, άρα πάμε στην 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΑΕ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147, υπέρ, κατά, αποχές,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 κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 θα ελέγξω την 158. 158. This is where some groups swap sides again. Uh, no. Yes. 23 υπέρ, 19 κατά. Um, recital. Μια ομάδα που αλλάζει. 159 υπέρ. Κατά. Δεν καταλαβαίνω να ελέγξουμε την 159. Um. and that's rejected. Απορρίπτεται. Κάπου να σηκώνετε και τα χέρια σας. Μάλλον είναι δύσκολο. 160 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται άρα σε ελέγξουμε δύο τις έκανα λάθος Κάποιος έχει μπει στον κόπο να καταθέσει μια τροπολογία και την ψηφίζουμε. Απορρίπτεται 24 κατά, 21 υπέρ, 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 160 καταπίπτει αν υιοθετηθούν όλες αυτές. 163 εγκρίθηκε, άρα 162 καταπίπτει. 164 καταπίπτει. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 είναι μετά, γιατί απορρίφθηκαν οι άλλες. 168 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε. 170. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται 27 υπέρ 19 κατά. Σωστά.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 που έχει καταπέσει επειδή ε, υιοθετήσαμε, εγκρίναμε την... Τι γίνεται με την 174 και 175 καταπέφτουν και αυτές ή ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 κατά πίπτη 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 καταπίπτει 189 καταπίπτει 11 καταπίπτει πάμε στη 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 38 υπέρ, 5 κατά, 5 κατά, 3 αποχές. Τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα υπέρ, κατά και αποχές. Άλλοι δύο να ψηφίσουν, πέρα της ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 5 κατά, και τέσσερις αποχές. Ωραία. Αυτό ήτανε. Δεν έχουμε τελειώσει όμως, γιατί τώρα έχουμε και το άλλο κομμάτι που είναι η οδηγία. Μια μικρή λίστα ψηφοφοριών. Συμβιβασμός α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 2 υπέρ, Περιμένω το Ζαν Πολ. Τροπολογία 2 για την οδηγία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός B υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμό C υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο κείμενο ως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία 39 υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές. Και για το νομοθετικό ψήφισμα... Άλλοι τρεις να ψηφίσουν. Άλλος ένας. Πέρας. 38 υπέρ, 3 κατά, 4 εποχές. Μην χειροκροτείτε. Μπράβο, μπράβο, Λεωνάρντο. Okay. Um, uh, I've... Leonardo, do you want to uh, take the floor? Leonardo, Θέλεις ε, να πάρεις το λόγο για να μας πεις αν θέλεις να ξεκινήσεις διαπραγματεύσεις την πρώτη ανάγνωση. Ναι, Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους κοιόδης εισηγητές καθώς και τους βοηθούς τους. Θα ήθελα να κάνω μια δική μνήμα του συναδέλφου Μίγκελ Πόρτα. Το ξεκινήσαμε μαζί, αλλά δεν μπορέσαμε να περατώσουμε αυτή την εργασία. Και ευχαριστίε στην Γραμματεία, στην Κλέρ και τον Φρανσουά για την υπομονή τους και τι ικανότητε του. Βεβαίω, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι αυτά που κάναμε είναι ήδη κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ακολουθήσουμε την συνηθισμένη διαδικασία και θα συμπεριλάβουμε έναν εισηγητή και ένα σκιώδη εισηγητή. Η εντολή είναι η, η έκθεση που ήδη ψηφίσαμε και ο συνήθως θα αναφερθούμε στην Επιτροπή και θα συντονίσουμε ε, και θα το συντονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στο σημείο 14. Σημείο 14, Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Επιτροπή Προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα. Οπίνε. Τρία υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Περνάμε στο 2. επιτροπή Απασχόλησης. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός, Επιτροπή Προϋπολογισμού 4 απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμού 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. απασχόληση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμ... Από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Λέει δεν είναι συμβατός. Τροπολογία 4, συμβατή. Η 4 από την Επιτροπή Επασχόληση. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή επασχόληση 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για, να δούμε. Δεν δε σας είδα, δεν σας είδα. Ωραία, ψηφίσω. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 25-18. Συμβιβασμός 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός C σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. άλδιψε ε, ε, υπέρ, κατά, αποχιές ωραία, εγκρίνεται. Ωραία. Συνεχίζουμε στο D. Από την τροπή απασχόληση 6 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε, D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Περιορισμού 12 υπέρ κατά 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμού 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεν είναι συμβατή τροπολογία 5 Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη 5 καταπίπτει, περνάμε στη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από την Επιτροπή Πασχόλης 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από την Επιτροπή Πασχόλης 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε, ή υπερκατά, αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 Υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F υπέρ αποχές εγκρίνεται η 24 καταπίπτει, συμβασμό G, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, από την Επιτροπή Επασχόλησης 10, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά, από την Επιτροπή Προπολογισμού υπέρ κατά αποχές μισό λεπτό. Επιτροπή Προπολογισμού, η 18. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 30, 12, συμβιβασμός α πρώτο μέρος, ψερ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ΆΙΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα την προφορική τροπολογία του e προφορική τροπολογία ψήφι πέρα κατά αποχές για να δούμε, για να το ελέγξουμε Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίες Απορρίπτεται 21 υπέρ, 22 κατά. Μία δεύτερη προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ, ψήφι κατά. Αποχές. Μισό λεπτό γιατί δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει με το ΕΛΚ. Είστε υπέρ. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 18 κατά. Περνάμε τώρα στην 29, τροπολογία 29, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 20 υπερκατά που συγκρίνεται, προφορική τροπολογία D, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθυμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από την Επιτροπή απασχόληση 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, προϋπολογισμού 21 υπερκαταποχές εγκρίνεται προϋπολογισμού 22 υπερκαταποχές εγκρίνεται από την προϋπολογισμού 23 υπερκαταποχές εγκρίνεται συμβιβασμός J υπερκαταποχές εγκρίνεται 24 από την προϋπολογισμού Προπολογισμού εγκρίνεται 33 υπέρ αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση υπέρ, 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε το 15 λίγο ψηφίσετε. 24 υπέρ, 19 κατά, 16 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε λίγο 21 για να ελέγξουμε Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 23, 24 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές για να ελέγξουμε το 24. Δύο ακόμα. Εντάξει, έκλεισε η ψηφοφορία. 23 υπέρ 20 κατά 25 από την Επιτροπή Επασχόληση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογή 23 υπέρ κατά απορρίπτεται 40 υπέρκατα, κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 αμισό λεπτό, τον ελέγξω του 41. δύσκολο μου φαίνεται. Εγκρίνεται. Από την Επιτροπή επασχόληση 28 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από την Επιτροπή επασχόληση, 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σηκώστε τα χέρια σας. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Απασχόλησης 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ Τι είναι αυτό που... Για να δοκιμάσουμε. 34 υπέρ, κατά. αποχίες απορρίπτεται. Για να το ελέγξουμε. τέταρτο πάλι. obscuring Ola, so I can't see what you're doing. Um, uh, employment 35. Επιτροπή Απασχόληση 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από την Επιτροπή Απασχόλησης 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τελευταία σελίδα. Επιτροπή απασχόληση, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από την Επιτροπή Επασχόλησης 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε για το κείμενο πως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά κανένας 43 Κανένας δεν δεν κατά, δεν απήχε. Α, τη συνηθίσαμε την ομοφωνία εδώ. Ωραία, ωραία. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Για πιέστε τα κουμπιά. Ελάτε. Ελάτε. Τέσσερις ακόμα μας έμειναν. Τρεις που ανθίστανται στην ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 40 υπέρ, κανένας κατά. Η συγκητή θέλει να πάρει το λόγο σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία ή την πρώτη ανάγνωση. Yeah, I can there will be a... Ναι, ναι, επιβεβαιώνω ότι θα υπάρξει πρώτη ανάγνωση. Ως συνήθως η σύνθεση της ομάδας διαπραγμάτευσης θα είναι πρόεδρος, εισηγητής και σκιώδης εισηγητής. Ε, θα αναφερθούμε και πάλι στους συντονιστές και στην Επιτροπή όπως κάνουμε συνήθως. Θέλω να γνωρίζω. Όταν είχε όταν, έχει, όταν λαμβάνουν χώρα δέκα τριμερεί συζητήσει ε, οι δέκα είναι δωρεάν. Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι για λίγο δεν θα πω πολλά. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Α, οικονομικές καταστάσεις, μάλιστα. Πρόκειται για την έκθεση γνωμοδότηση συγκεκριμένα του Βολφ Κλίντ. Τροπολογία 1 ψήφι υπέρ. Α, όχι, έχει αποσυρθεί, εντάξει. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Ναι, Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά. Να ελέγξω παρακαλώ 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 18 προς 21. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται νομίζω με την ίδια διαφορά ψήφων. Αλλά να ελέγξουμε, εντάξει. Εγκρίνεται. Τώρα δεν θυμάμαι. Ε, μήπως κλείσαμε πολύ νωρίς την ψηφοφορία. Μήπως καλό θα ήταν να ξαναψηφίσουμε γιατί ενώ δεν είχαν ψηφίσει τρεις κλείσαμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε. Okay. Keep on voting. Everybody press. Ψηφίστε παρακαλώ. Δύο ακόμη έχουμε. Δεν έχουν ψηφίσει, μήπως δεν θέλουν, δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, τώρα κλείνουμε. Ξεκολουθεί να εγκρίνεται με διαφορά μιας ψήφου. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Σοσιαλιστές να σκόνουν τα χέρια τους παρακαλώ. Πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχω την 52. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές. Abstentions. Απορρίπτεται. Καλώς να ελέγξω. Ελέγχουμε λοιπόν την 54. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται 17 υπέρ 22 κατά. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11 υπέρ, 25 κατά. 59 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ όχι έχει καταπέσει 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 όχι. 77 καταπίπτει όχι εντάξει. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Γ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ε, θεωρώ καλύτερο να ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 18 υπέρ 20 κατά. Πού πηγαίνουμε τώρα. Συμβαστική δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117 υπέρ, κατά, αποχές. Η ομάδα ECR τι κάνει, δεν βλέπω. 117 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. 117. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120. Μισό λεπτό ήταν το ίδιο, ναι. Συμβαστική εύσηγμα τα αφιπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 140. Υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 140. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 141. Όχι, είναι ταυτόσιμο. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική GZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ. Όχι. Όχι πίπτη. Πάμε στην 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. «176 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική H. τα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές 26 πρέπει να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 27 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά αποχές δεν έχω καταλάβει τι έχουν ψηφίσει οι σοσιαλιστές, να ελέγξουμε την 31. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 19 υπέρ 20 κατά. Συμβιβαστική I ή θ. Εγκρίνεται. J, J υπέρ κατά αποχής Εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 35 υπέρ, 4 αποχές, κανείς κατά. Άρα συγχαίρουμε τον Βόλφ. Χαίρομαι γιατί δεν θα πάμε σε τριμερή διάλογο. Έχουμε άλλη μια ψηφοφορία. Thank you. Okay. So this is... Λοιπόν, νομοδότηση τη ΣΥΡΠΑ, τι είναι, τη διαφάνεια. Λοιπόν, φύγαμε. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται.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 Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 17 υπέρ 20 κατά. 45 τροπολογία. Μαζί με τις 46 και τις 47. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, όχι, καταπίπτει. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 μαζί με 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτονται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60. Έχουμε προφορική τροπολογία που αντικαθιστά τις αναφορές στο platform σε, με access point. Ποιοι είναι υπέρ της, της προφορικής τροπολογίας υπέρ. Κατά, πόχες, εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται 62 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται 63. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται Συμβαστική Σ, Γ, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, Οι σοσιαλιστές τι ψηφίζουν. Είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν. Ψηφίζουμε τώρα το συνολικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 34 ψήφοι πέρ, μία κατά, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Στα διάφορα δεν έχουμε κάτι. Επόμενη συνεδρίαση λοιπόν Δευτέρα 25 Ιουνίου. Ευχαριστώ όλες και όλους.